Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε την απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα φροντίσουμε να μην υπάρξουν προβλήματα χρόνου στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας ε, σκεφτήκαμε χρήσιμο και για τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας αλλά και για τους ευρωβουλευτές γενικά να παρακολουθήσουμε μια γενική παρουσίαση της ε, μεταρρύθμισης της κοινή αγροτικής πολιτικής που ολοκληρώθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους. Συζητήσαμε ε, για το θέμα αυτό με τον Επίτροπο Τσιόλος και με το Γενικό Διευθυντή της, Επιτρο... της ε, Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πλέβα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ε, θετικά και μας διαβεβαίωσαν ότι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη Γεωργίας θα ετοιμάσει μια διεξοδική παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα είχαμε ήδη μια πρώτη περίοδο εφαρμογής της ΚΑΠ, οπότε η παρουσίαση θα είναι εμπλουτισμένη και με τις καινούργιες εμπειρίες. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η παρουσίαση, αυτό το σεμινάριο και για τους παλιότερους βουλευτές, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και ιδιαίτερα και για τους εισηγητές της μεταρρύθμισης, τον κύριο Νταντέν, τον κύριο Καπόλα Σάντος, και σίγουρα και οι εισηγητές θα λάβουν μέρος στη συζήτηση. Επίσης, καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Έχουμε εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας σε υψηλότερο επίπεδο. Έχουμε το Γενικό Διευθυντή Γεζή Μπόγκταν Πλέβα. Και με βάση το πρόγραμμα που λάβατε θα περάσουμε στο σεμινάριο. Πρώτα θα ακούσουμε μία εισαγωγή από το Γενικό Διευθυντή Μπόγκταν Πλέβα. ο οποίος όμως ε, λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων θα φύγει αμέσως μετά την παρουσίασή του. Θα ακούσουμε όμως στη συνέχεια ειδικέ παρουσιάσεις από διευθυντές ε, της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη και θα έχουμε και γύρω έρωτα απαντήσεων μετά τις επιμέρους παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τη Γενική Διευθύνση Άγκρη Γεωργίας για την αποδοχή της πρότασης και για τη διοργάνωση του σεμιναρίου. Και θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Γέζη Μπόγκταν Πλέβα, το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Και κατόπιν βάσει το πρόγραμμα που έχουμε μοιράσει, θα ακούσουμε τις επιμέρους παρουσιάσεις των διευθυντών. Κύριε Πλέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερος που σήμερα μαζί με τους συναδέλφους θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα κύρια στοιχεία της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής και τις προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της. Από τη δεκαετία του 90, η κοινή αγροτική πολιτική παρουσίασε σημαντικές αλλαγές. Από προστασία των συνόρων, εξαγωγικές επιστροφές, τιμές παρέμβασης, περάσαμε σταδιακά από ένα σύστημα εναυσμάτων για το πόσο και πώς παράγει ο Γιώργος σε ένα σύστημα που περιστρέφεται γύρω από το τρόπο και από το λόγο παραγωγής. Περάσαμε από το τι στο πόσο και στο γιατί. Η κοινή αγροτική πολιτική βοήθησε τους γεωργούς να ανταποκριθούν καλύτερα στα, στις ανάγκες της αγοράς και να εντάξουν τη γεωργία στην γενική οικονομία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ε, στήριξης της, πολιτικής, της αγροτικής πολιτικής. Προσπαθήσαμε λοιπόν να προσαρμόσουμε την, αγροτική, την κοινή αγροτική πολιτική στις, ε, στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, το οποίο και έλαβε την τελική απόφαση. Αυτό το χαρακτήρα είχαν ε, οι διαβουλεύσεις και η διαδικασία διαβουλεύσεων στο παρελθόν. Στο παρελθόν ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδινε τη γνώμη του. Έδινε γνωμοδότηση που είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά η λήψη υπόψη της δεν ήταν υποχρεωτική. Με τις πρόσφατες όμως μεταρρυθμίσεις της κοινή αγροτικής πολιτικής, τα πράγματα άλλαξαν. Το θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε. Από το 2010, με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, η, κανονιστική, η νέα κανονιστική διαδικασία έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων για την κοινή αγροτική πολιτική άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού και αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και στο διαδικαστικό της σκέλος, γιατί έχουμε πια μια πιο περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία λήψη αποφάσεων, αλλά επηρέασαν και την ουσία οι αλλαγέ, την τελική έκβαση δηλαδή και την τελική διαμόρφωση της ΚΑΠ. Η αλλαγή της πολιτικής έλαβε χώρα στο πλαίσιο της συζήτησης ε, για το γενικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινής αγροτικής πολιτικής, ο προϋπολογισμός μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης με βάση τις σταθερές τιμές. Και μάλιστα βλέπετε ε, τις γεωργικές δαπάνες με τρέχουσες τιμές από τους πίνακες. Από το 2014 μέχρι το 2020 έχουμε σταθερές δαπάνες ανά έτος. Με την τρέχουσα όμως οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, οι οικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να δίνουν στήριξη σε μια φιλόδοξη αγροτική πολιτική που ανταποκρίνεται στο 37,8% του συνόλου των κοινοτικών δαπανών για την περίοδο 2014-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διεξοδικό έλεγχο του υφισταμένου πλαισίου πολιτικής και προσπάθησε να το προσαρμόσει στις περιβαλλοντικές, ε, εδαφικές και άλλες ανάγκες που θα αντιμετωπίσει η Γεωργία. Στην ανάλυση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε τρεις πρωταρχικούς στόχους. Την ανάγκη προώθησης της ασφάλειας των τροφίμων, βοηθώντας τον κλάδο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ε, που δημιουργεί ε, η αστάθεια και η αβεβαιότητα στις αγορές και η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Δεύτερον, εξασφάλιση της ε, μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, βάζοντας τις κλιματικές δράσεις και την ε, βιώσιμη διαχείριση των πόρων ε, στο επίκεντρο της δράσης μας. Και τρίτον, συμβολή στις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις τεσσάρων τομέων διαφυλάσσοντας ε, τη διαρθρωτική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς, τροποποιώντας τα τέσσερι βασικού τέσσερις βασικούς μηχανισμούς της κοινή γεωργική πολιτικής, Τι άμεσε ενισχύσει, την κοινή οργάνωση αγοράς, την αγροτική ανάπτυξη και την πολιτική ανάπτυξη τη υπαίθρου. Οι συνάδελφοι θα σας περιγράψουν διεξοδικά τους μηχανισμούς αυτούς και επίσης το τέταρτο ήταν οριζόντιος κανονισμός. Ακροθυγώς θα σας παρουσιάσω μερικά μόνο στοιχεία της μεταρρύθμισης. Για τις άμεσες ενισχύσεις. Οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να αποτελούν το κυριότερο μέσο της πολιτικής από οικονομική άποψη γιατί αντιστοιχούν στο 80% του προϋπολογισμού της κοινή αγροτικής πολιτικής. Οι άμεσες ενισχύσεις θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων παρέχοντας μια αξιόπιστη πηγή εισοδήματο για τους παραγωγούς. Με την τελευταία μεταρρύθμιση Περάσαμε από το σύστημα ιστορικών πληρωμών με σύστημα αναφοράς σε ένα σύστημα επιδοτήσεων αναέκταση. Έχουμε πιο ισότιμη μεταχείριση των γεωργών άσχετα από τις ιστορικές επιλογές παραγωγής τους. Η νέα διαμόρφωση του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων στηρίζεται σε κάποια υποχρεωτικά καθεστώτα. Το νέο ε, καθεστώς βασικής πληρωμής, τις ε, νέες ενισχύσεις για τους ε, νέους, νέους ερχόμενους γεωργούς και τους, τις πράσινες ενισχύσεις, τις πράσινες πληρωμές. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι υποχρεωτικά για όλα τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη έχουν την ευκαιρία ένα τμήμα των άμεσων ενισχύσεων να να το διοχετεύσουν σε άλλους δικαιούχους, ε, σε τομείς ή σε περιοχές ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που εντοπίζουν. Και αυτό γίνεται εθελοντικά. Πρόκειται για την εθελοντική συνδεδεμένη ενίσχυση, την ενίσχυση περιοχών με εδαφικούς περιορισμούς και την αναδιανεμητική ενίσχυση. Εδώ ισχύει προαιρετικό σύστημα. Τα κράτη-μέλη επίση ε, και εθελώ μπορούν να εφαρμόσουν και το καθεστώ για του μικρού καλλιεργητέ. Με τις αλλαγές ε, στην κοινή οργάνωση αγοράς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον γεωργικό τομέα. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την άρση των περιορισμών στην παραγωγή, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας διευρυμένο και ένα τρόπο διαχείρισης των κρίσεων. Οι περισσότερες ποσοστώσεις έχουν καταργηθεί ή θα καταργηθούν ως νούπο. Οπότε οι παραγωγοί μπορούν να αποφασίσουν με βάση τα σημάδια που παίρνουν από την αγορά, με βάση τις ανάγκες της αγοράς, πότε και πόσο να παράγουν. Τα νέα μέσα της πολιτικής αφορά, αφορούν και τη λειτουργία της αλυσίδας ανεφοδιασμού. Εδώ ενισχύουμε το πλαίσιο για τις ενώσεις παραγωγών, τους συνεταιρισμούς τους και τις διακλαδικές οργανώσεις. Τέλος, θα αναφερθώ στην αγροτική ανάπτυξη που είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Η νέα κοινή για αγροτική πολιτική θέτει την αγροτική ανάπτυξη στο επίκεντρο, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής και επικεντρώνεται σε στρατηγικούς στόχους αλλά και σε στοχευμένες πρωτοβουλίες. Η αγροτική ανάπτυξη είναι θεμέλιο της γεωργίας. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα συνεχίσουν να, καταρτίζουν τα πολιετή τους προγράμματα με βάση τα τα μέτρα και τα κονδύλια τους ε, και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών. Πάντως, η νέα πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα είναι πιο ολοκληρωμένη και θα συνδυάζεται με τα διαρθρωτικά ταμεία και το επενδυτικό ταμείο. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο εναρμόνισης όλων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου και χάρη στην εναρμόνιση αυτή θα βελτιωθεί ο προγραμματισμός και θα αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των περιφερειών ενώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Όλα αυτά θα γίνουν μέσω της Εθνικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με πολλές αρμόδιες αρχές, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία συνολική συνεκτική στρατηγική. Συνεχίζονται τώρα οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη επί των συγκεκριμένων προτάσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Σε αυτή τη σύντομη εισαγωγή θα ήθελα να σας πω ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήταν η πρώτη εμπειρία συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Μείναμε ικανοποιημένοι από αυτή την πρώτη εμπειρία και συνεργασία. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι στο μέλλον μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Πιστεύω επίσης ότι με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τώρα σχηματίζεται θα εντατικοποιηθεί ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μελλοντικέ προκλήσεις του γεωργικού μας κλάδου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πλέβα, κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσίαση και ευχαριστούμε που ήρθατε στο σεμινάριο. Περνάμε τώρα στις επόμενες παρουσιάσεις με βάση το πρόγραμμα που έχετε λάβει. Θα ακούσουμε την παρουσίαση για τις άμεσες ενισχύσεις. Θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή κύριο Πιέρ Μπασκού που θα μας κάνει την ενημέρωση για το θέμα αυτό. Κατόπιν θα έχουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω λοιπόν με την παρουσίαση αυτή. L'objet de cette présentation est de donner un bref aperçu. Προσπαθήσω σύντομα να σας παρουσιάσω το νέο σύστημα άμεσων πληρωμών. Ένα νέο σύστημα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από το 2015 για τα επόμενα έξι χρόνια. Να σας θυμίσω τους βασικούς στόχους αυτού του νέου μέσου. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο είναι ήδη υπάρχον και δείχνοντάς σας και τις πιο πιθανές αλλαγές, βασικές αλλαγές σε επίπεδο εξωτερικών συγκλήσεων, σε επίπεδο νέων αρχιτεκτονικών μορφών των άμεσων πληρωμών ή ενισχύσεων, επιμένοντας σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σε εισαγωγικά πρασίνισμα της μεταρρύθμισης αυτής. Λίγα λόγια τώρα για τα μέσα τα νέα αυτής της μεταρρύθμισης. Υπάρχει ένα νέο σύστημα λοιπόν άμεσων ενισχύσεων. Τρεις στόχοι. Πρώτος στόχος είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα. Η διασφάλιση συνεπώς της προμήθειας τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενίσχυση των εισοδημάτων και σε επίπεδο άμεσων ε, εισοδημάτων και σε επίπεδο σταθερότητας των εισοδημάτων αυτών, βελτίωση της αϊφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, σαφής αναγνώριση του σημαντικού ρόλου των γεωργών ως παραγωγών ιδιωτικών αγαθών, αλλά ταυτόχρονα και παροχέων περιβαλλοντικών αγαθών, ιδιαιτέρως μέσω της στήριξης η οποία χορηγείται προς τους γεωργούς και μέσω καλλιεργιών και μορφών καλλιέργειας ε, συμβατών με τις κλιματολογικές αλλαγές. Και τρίτος στόχος θα έλεγα αυτού του νέου συστήματος άμεσων ενισχύσεων είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω της σωστής στήριξης σε συγκεκριμένες περιοχές έτσι ώστε να διατηρήσουμε και γιατί όχι να αναπτύξουμε ε, την οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική, ε, γενικά και την οικονομία των ε, περιοχών αυτών της υπαίθρου. Το σύστημα θα είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτα θα στοχεύουμε καλύτερα. Οι άμεσες ενισχύσεις δηλαδή θα στοχεύουν ε, ακριβώς με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των δραστήριων γεωργών αποκλείοντας όλους όσους έχουν περιθωριακή σχέση με το γεωργικό τομέα, στοχεύοντας σωστά τις ανάγκες των νέων γεωργών και στοχεύοντας σωστά ε, τις ανάγκες ορισμένων τομέων και ορισμένων περιοχών και ορισμένων μορφών εκμετάλλευσης ανάλογα με το μέγεθός τους. Και αναφέρομαι εδώ στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις γεωργικές ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα μέσω μιας πιο δίκαιης κατανομής των επιδοτήσεων, μέσω της σύγκλησης σε επίπεδο δημοσίας επιδότησης, η λεγόμενη δηλαδή εξωτερική σύγκληση και στο εσωτερικό των κρατών μελών η λεγόμενη εσωτερική στήριξη. Δυνατότητα επίσης και χρήσης του μέσου του αναδιανεμητικού έτσι ώστε να υπάρξει σωστή κατανομή ανάμεσα στις εκμεταλλεύσεις διαφορετικού μεγέθους. Και ένας τρίτος ε, θα έλεγα στόχος είναι οι λεγόμενες πράσινες πληρωμές οι οποίες θα ακολουθηθούν από μια απλούστευση αλλά και ενίσχυση του συστήματος της αιρεσιμότητας Ερεσιμότητα τι είναι, είναι αυτό που συνδέει τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων με άλλες μορφές επιδοτήσεων που σέβονται βέβαια την κοινοτική νομοθεσία. Ένα σύστημα δηλαδή ερεσιμότητας το οποίο θα έχει λιγότερες νομικές δεσμευτικές διατάξεις αλλά θα επηρεάζει πολύ πιο ισχυρά το γεωργικό τομέα και θα επηρεάζει επίσης πιο ισχυρά προς την καλή κατεύθυνση το περιβάλλον. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα έχει σαν στόχο να αντικατοπτρίζει σωστά ε, τις αποφάσεις οι οποίες έχουν ε, ληφθεί σε επίπεδο εξωτερικών μορφών σύγκλησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης για το 2020 επί τη βάση των άμεσων ενισχύσεων όπως υπάρχουν σήμερα αναμονάδα. Βλέπετε λοιπόν το αριστερό τμήμα ε, της κάθε στήλη αφορά την σημερινή κατάσταση και το δεξί τμήμα, τη δεξιά στήλη, μπλε αν τη βλέπετε έτσι εσείς, που αφορά την λεγόμενη εξωτερική σύγκληση και βλέπουμε μια γυθνίαση ανάμεσα σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα ανάμεσα σε χώρες που βρίσκονται στα δύο άκρα αυτού του γραφήματος. Δηλαδή και ε, επιδοτήσεις εθνικές και άμεσες πληρωμές στον ορίζοντα του 2020. Τώρα για τη νέα αρχιτεκτονική των άμεσων πληρωμών. Εδώ έχουμε διαφορετικές, διαφορετική διαστρωμάτωση σε σχέση ε, με τις συνδεδεμένες και ε, αποσυνδεδεμένες πληρωμές. Από το 2015 θα έχουμε έξι διαφορετικά καθεστώτα. Τρία θα είναι υποχρεωτικά και τρία εθελοντικά. Τα υποχρεωτικά αφορούν τις βασικές πληρωμές, τις πληρωμές βάσης, το ενιαίο σύστημα πληρωμών για επιφάνειες και ε, αυτό με την εξαίρεση βέβαια των συνδεδεμένων πληρωμών. Δεύτερο καθεστώς υποχρεωτικό είναι οι λεγόμενες πράσινες πληρωμές και τρίτον είναι η ειδική αντιμετώπιση, το ειδικό μέσο για τους νέους γεωργούς. Ε, βλέπετε επίσης και τα τρία γκρίζα σε εισαγωγικά εθελοντικά καθεστώτα. Πρώτον, το σύστημα των συνδεδεμένων πληρωμών που επιτρέπει σε επίπεδο επιδοτήσεων κρατικών κατελάχιστον βοήθεια σε, ορισμένες, σε ορισμένους τομείς οι οποίοι θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικοί ε, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Ένα δεύτερο εθελοντικό καθεστώς είναι το σύστημα των άμεσων επιδοτήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές με εγγενείς φυσικές δυσκολίες. Και τέλος έχετε το μέσο αναδιανομής το οποίο επιτρέπει την στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Βλέπετε λοιπόν κάποιες πιο συγκεκριμένες εδώ ρυθμίσεις που ισχύουν για το κάθε ένα από αυτά τα καθεστώτα, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην παρούσα φάση. Πάντως, τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να εισάγουν ένα ειδικό καθεστώς για τους μικρούς γεωργούς επί εθελοντικής βάσεως. Πρόκειται για ένα σύστημα απλουστευμένο σε επίπεδο διαχείρισης, απλουστευμένο σε επίπεδο ελέγχου και που ε, νομίζω θα ωφελήσει τους γεωργούς. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο είναι το πιο καινοτόμο της μεταρρύθμισης αυτής, είναι η εισαγωγή ε, του λεγόμενου πράσιν, της λεγόμενης πράσινης πληρωμής, δηλαδή κάτι το οποίο έρχεται σε αντιστάθμιση, αν θέλετε, ε, της χρήσης ορισμένων καλλιεργητικών πρακτικών ευεργετικών για το περιβάλλον. Ε, υψηλή δημοσιονομική επιβάρυνση 30% των εθνικών φακέλων που ε, βασίζονται ε, στις, ε, που περνούν μέσα από τις έμεσες ενισχύσεις. Λοιπόν, αν αυτή η άμεση πράσινη ενίσχυση είναι ένα βασικό, αν θέλετε, χαρακτηριστικό του πρασινίσματος, επαναλαμβάνω εισαγωγικά της ΚΑΠ, αυτό είναι κάτι που εντάσσεται γενικότερα στην πολιτική μας για την ΚΑΠ. Βασίζεται στην στον μηχανισμό αιρεσιμότητας που συνδέει τη δημόσια επιδότηση με το σεβασμό μεταξύ άλλων και του περιβάλλοντος, των κανόνων για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρία μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν υποχρεωτικά στον πρώτο πυλώνα. Καταρχάς ε, μέτρα που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, και μέτρα τα οποία στην παρούσα φάση δεν είναι δεσμευτικά επί τη βάση αυτών των δύο τμήματων, ερεσιμότητα και πράσινες πληρωμές, έχετε και το τρίτο συστατικό εδώ, το οποίο είναι τα μέτρα, τα περιβαλλοντικά για την ανάπτυξη της υπαίθρου, που είναι μέτρα εθελοντικά, πλέον στοχευμένα και τα οποία επιτρέπουν να ανταποκριθούμε σε πιο συγκεκριμένους στόχους και ερωτηματικά τοπικά. Αυτά τα τρία συστήματα, αυτά τα τρία πεδία αν θέλετε πρασινίσματος της κοινή αγροτικής πολιτικής συμπληρώνονται από τι άλλο μπορεί να γίνει στον τομέα της έρευνας και των νέων συστημάτων χορήγησης συμβουλών στην γεωργική δραστηριότητα. Κάποιες λεπτομέρειες τώρα για τα τρία μέτρα πρασινίσματος εισαγωγικά επαναλαμβάνω. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν από τους γεωργούς για να πάρουν αυτή την πληρωμή, καταρχάς ε, ε, μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων ε, για την συγκράτηση των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το σύνολο, συγκεκριμένα ποσοστά σε σχέση με το σύνολο της εκμετάλλευσης, ανάλογα αναπεριοχή το οποίο θα αποτρέψει τη μετατροπή της χρήσης των γεών. Δεύτερον, ε, πολλαπλές καλλιέργειες που βοηθούν την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα των υδάτινων πόρων με δύο ή τρεις ε, ε, καλλιέργειες διαφορετικές σε μία επιφάνεια. Και το τρίτο μέτρο είναι οι επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος. Εδώ η υποχρεωτική λήψη υπόψη τους θα πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 5% του συνόλου των επιφανειών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη της βιοπικιλότητας στον γεωργικό τομέα και να δώσουν την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να καθορίσουν και να δημιουργήσουν μια δεσμευτική ρύθμιση μέσω της επιλογής περισσότερων 10 τύπων επιφανειών. χρησιμοποιούμε αγγλικά αρχικά εδώ και έχετε διαφορετικές ονομασίες για τις εκμεταλλεύσεις αυτές. Για τα EFA, εν πάση περιπτώσει, μέσω τοπιογραφικών, μέσω ε, ε καλλιεργιών ειδών φυτών πλούσιων σε άζωτο κτλ. Όλα αυτά δίνουν την δυνατότητα στα κράτη-μέλη εφόσον το επιθυμούν να δημιουργήσουν και ένα σύστημα ισοτιμιών το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων πρασινίσματος και σε επίπεδο οικολογικό στο δεύτερο πυλώνα, εξίσου φιλόδοξων οικονομικά και οικολογικά ή μέσω και των, συστημάτων, των λεγόμενων συστημάτων πιστοποίησης. Τώρα για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του συνόλου αυτών των άμεσων ενισχύσεων. Πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Η υγιής οικονομική διαχείριση του συστήματος και είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα θα συνεχίσει να βασίζεται στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και ιδιαίτερα στο σύστημα ταυτοποίησης και ανείχνευσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιφανειών που επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή αυτών των άμεσων ενισχύσεων. Δύο στοιχεία τώρα τα οποία είναι σημαντικό να σημειωθούν εδώ σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις. Το πρώτο έχει σχέση με τις γεωχωρικές σε εισαγωγικά πάντα ρυθμίσεις τεχνολογικά που θα καταστήσουν τη διαχείριση του συστήματος πολύ πιο αποτελεσματική και εύκολη. Και δεύτερον η εισαγωγή ειδικών στρωμάτων στο σύστημα εντοπισμού των γεωργικών εδαφών σχετικών με το πρασίνισμα και σχετικών με τις επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος, τα στρώματα EFA στα αγγλικά. Κάτι το οποίο θα επιτρέψει την σωστή διαχείριση του συστήματος αυτού στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Κλείνοντας, να υπενθυμίσω ότι το νέο σύστημα άμεσων πληρωμών ενισχύσεων θα επιτρέψει στο μέλλον να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή της πολιτικής προς μια πιο αηφόρο γεωργική δραστηριότητα που θα επιτρέψει να ληφθούν υπόψη καλύτερα οι παράγοντες οι γεωοικονομικοί και γεωπολιτικοί. Μέσω και μιας μεγαλύτερης ευελιξίας που δίδουμε στα κρατη έτσι ώστε να προσαρμόζουν αυτό το νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων στα ειδικά τους χαρακτηριστικά. Τώρα για τις βραχυπρόθεσμες δραστηριδάσεις Εδώ και αρκετούς μήνες βέβαια και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα υπάρχει μια δραστηριότητα πολύ σημαντική εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος στα κράτη-μέλη με μια σημαντική υποστήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα φάση είμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης των γνωστοποιήσεων και των ανακοινώσεων που έγιναν από τα διάφορα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Δύο χρονικές προθεσμίες που πρέπει να, ε, να λάβουμε υπόψη μας εδώ. εξέταση των εμπειριών μετά από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ιδιαίτερα στον τομέα των άμεσων ενισχύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των διοικητικών επιβαρύνσεων, γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων και στην δημιουργία των ισότιμων ε, τρόπων αντιμετώπισης αυτών των διαχειριστικών προβλημάτων στις διάφορες χώρες. Και δεύτερη προθεσμία είναι ο Μάρτιος του 2017. Τότε θα υπάρξει μια νέα έκθεση για τις ευαίσθητες οικολογικά επιφάνειες οι θα μας δώσουν, η οποία έκθεση θα μας δώσει στοιχεία για τις νέες αυτές μεθόδου και θα προτείνουμε 5 ε, με 7% αύξηση περαιτέρω για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα βασικά στοιχεία ακριβώς αυτού του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, θα έχουμε τώρα ένα γύρο έρωτα απαντήσεων, αλλά παρακαλώ οι ερωτήσει να περιορίζονται στις άμεσες ενισχύσεις. Γιατί αργότερα θα μιλήσουμε για την αγροτική ανάπτυξη, τον οριζόντιο κανονισμό ή την κοινή οργάνωση αγοράς. Τώρα θα επικεντρωθούμε μόνο στις άμεσες ενισχύσεις. Παρακαλώ κάθε φορά οι ερωταπαντήσεις να περιορίζονται στο θέμα που μόλις πριν από λίγο ακούσαμε. Πρώτα ο κύριος Δεκάστρο. Γιατί αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή Πλέμπα. Έπρεπε να φύγω κάποια στιγμή, αλλά να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή Μπασκού και όλη την ομάδα της Επιτροπής που βλέπουμε εδώ σήμερα, μετά από την τεράστια προσπάθεια που κάναμε μαζί πάνω από 50 φορμές τριμερών διαλόγων μεταξύ μας. Για πρώτη φορά είναι πλάκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθεια αυτή ε, συναπόφασης. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπογραμμίζουμε και τον στόχο ακριβώς αυτού του σεμιναρίου, ε, το οποίο θα δείξει στους νέους βουλευτές την δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα και όπως υπόθηκε από τον Διευθυντή Πλέμπα στην αρχή, με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Επιτροπή αυτή έχει πραγματικά αλλάξει τις δραστηριότητές της κατά πολύ. Σήμερα έχουμε πλέον μια συγκεκριμένη σημαντικότατη ευθύνη γιατί η συναπόφαση δεν επιτρέπει πλέον να κάνουμε απλές ε, κρίσεις επί της ουσίας ίστο, αλλά να παίρνουμε αποφάσεις εκτελεστικές ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα. Τώρα, Ακούγοντας αυτά που είπατε για τις άμεσες ενισχύσεις, ε, πράγματι έρχονται στην επιφάνεια νομίζω κάποιες μορφές ανησυχίας. Δηλαδή κάναμε μια μεταρρύθμιση η οποία στα πλαίσια του λεγόμενου greening και στα πλαίσια της ερεσιμότητας ε, δίδει περισσότερο βάρος στο περιβάλλον. Υπάρχει μια υψηλότερη ευαισθησία θα έλεγα για το περιβάλλον. Και ιδιαίτερα η παρουσίαση του Διευθυντή Μπασκού δείχνει ότι είναι τόσο περίπλοκο το θέμα αυτό που δημιουργεί πρόβλημα και μας κάνει να ανησυχούμε. Καταρχάς να ανησυχούμε σε σχέση με τους γεωργούς, γιατί εμείς θέλαμε το πράγμα να είναι πολύ, λιγότερο, πολύ περισσότερο κατανοητό, πιο απλό που να τους διευκολύνει τη ζωή και την πρόσβαση στα βοηθήματα που παρέχει η ΚΑΠ. Δεύτερον, τα προβλήματα προέρχονται επίσης και από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να ελέγξουν τις εφαρμογές αυτές και θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τα ειδικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των κανόνων που διαφέρουν μεταξύ τους. Εγώ δεν θα μπω εδώ επί της ουσίας, αλλά θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε ένα χρόνο πριν από το greening, η δυνατότητα ελέγχου αξιολόγησης ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι ώστε να κάνουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις αν θέλετε, διορθώσεις αν επιθυμείτε, αν τυχόν αποδειχθεί το σύστημα αυτό περίπλοκο για τους γεωργούς αλλά και για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα αυτή και θα το ζητήσουμε σίγουρα από τον νέο Επίτροπο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Πλιουέλ και να πω ότι είναι πάρα πολύ, παραδοσ... πολύ παρα... ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Πολύ καλή η παρουσίαση και σας συγχαίρω λοιπόν. Αλλά φυσικά μας υπενθυμίζει πάρα πολλά από τις μακρές συναντήσεις που είχαμε πριν από κάποιο καιρό. Και πολλές από τα πολλά από τα ακρονίμια που τα είχα ξεχάσει, τα θυμήθηκα. Πάντα λοιπόν καλό είναι να μας τα υπενθυμίζετε αυτά. Αυτό που ήθελα να σας ε, πω σήμερα εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το εξής. Πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στους αγρότες για το τι πρέπει να κάνουν την επόμενη άνοιξη και δεν μπορούν να βρουν απαντήσεις και μου λένε ότι δεν τους δίνετε εσείς τις απαντήσεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το έργο σας, αλλά πρέπει εκ παραλίλου να σας πω ότι δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί τώρα Δεν θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να δούμε τι συζητάμε. Για παράδειγμα, η τομή οικολογικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για ερωτήσεις, τις οποίες χρειάζονται απαντήσεις οι άγροτες, γιατί οι αγρότες κατηγορούν τους τοπικούς ηθήνοντες και αυτοί στρέφονται σε εσά για απαντήσεις. Δεν μπορούν να απαντήσουν χωρίς εσάς. Η προσωπική μου λοιπόν εμπειρία είναι η εξή. Ό,τι ερμηνεία και να δίνετε στην εφαρμογή της νέας αυτής μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, μπορείτε να μας πείτε και να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα υπάρξει αναδρομική αλλαγή από το δικαστήριο όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Από το ελεγκτικό συνέδριο μάλλον. Λέγοντάς μας ότι η εφαρμογή έγινε με λάθος τρόπο παρά το γεγονός ότι ακολούθησαν την καθοδήγηση των Βρυξελών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί κοστίζει εκατομμύρια σε κάποιες περιφέρειες όταν αναδρομικά προσπαθούν να διορθώσουν τα σπασμένα. Θα πρέπει να σας πω με πάσα σαφήνεια ότι θεωρώ ότι είναι καλή η ευκαιρία να γίνει αυτό σήμερα θα πρέπει να αντιληφθείτε την ανησυχία που υπάρχει από αυτούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν όσα εμείς αποφασίσαμε πριν από κάποιους μήνες. Δεν μπορώ να σας το τονίσω επαρκώς. σε ό,τι αφορά τη, το πρασίνισμα αυτό και τη, τα προϊόντα αυτά που συμβάλλουν στο πρασίνισμα, εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ δυνατοί από την περιφερειά μου, αλλά ούτε πρόκειται να είναι αναδική αυτή η τάση, γιατί δεν έχουμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε στα ερωτήματά μας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να αναβάλουμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους μέχρι ότου να ξέρουμε συγκεκριμένα τι συζητάμε. Ευχαριστώ. Κύριος Ντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρουσιάσεις, αλλά εγώ έχω σοκαριστεί από το αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτής, ακόμα και με τη διαδικασία της συναπόφασης, γιατί εξ αρχής είχα προειδοποιήσει και ούτε καν στην ομάδα μου δεν είχαμε πλειοψηφία. Αυτό το πράσινισμα, το πρασίνισμα στην πρώτο πυλώνα θα κατέληγε σε γραφειοκρατικό και βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος ε, κατάρτισης και η κοινή αγροτική πολιτική τέθηκε σε εφαρμογή. Αυτό που έχουμε μπροστά μας ε, είναι το πιο φρικτό και πιο γραφειοκρατικό πράγμα που έχει καταλήξει ποτέ μπροστά μας. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται στο πρώτο πυλώνα, πόσο χατιά έχουμε. Όποιος τα καταφέρει να τα διαβάσει θα καταλήξει τρολοκομείο. Εγώ χαίρομαι που ο Επίτροπος Τσιόλος δεν θα είναι εδώ τα επόμενα πέντε χρόνια γιατί ήταν ο χειρότερος δυνατός ε, ε, Επίτροπος στην Ευρώπη από τότε που υπάρχει γεωργική πολιτική. Και ελπίζω να μην αναλάβει κανείς ε, από τους προηγούμενους γιατί όλοι συνυπεύθυνοι είναι. Κοιτώντας λοιπόν τι λέει το κείμενο. Πώς ένας αγρότης να τα εφαρμόσει αυτά τα προγράμματα είναι απολύτως απαράδεκτο και αδύνατο για το πρασίνισμα το 2016 σε ό,τι αφορά την αναβολή. Ήξερα ότι δεν είναι έτοιμες οι προδιαγραφές, αλλά ακόμα και στην Επιτροπή Γεωργίας τελικά δεν ε, πέρασε η άποψή μου αυτή. Ήταν προβλεπόμενο ότι οι εκτελεστικοί κανονισμοί δεν επρόκειτο να είναι έτοιμοι. Και τα γραφεία μας ε, βομβαρδίζονται από τηλεφωνήματα γιατί οι αγρότες τώρα κάνουν την, ε, την εμπορνή εισοδιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς θα εφαρμόσουν όλα αυτά τα μέτρα για το πρασίνισμα. Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε λοιπόν τους γεωργούς αυτούς και κάποιος είπε ότι δίνουμε 6 δισεκατομμύρια στους ε, αγρότες και τι αποκομίζουμε τελικά από αυτό. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ακόμα πιο ακριβό είναι πραγματικά απαράδεκτη η κατάσταση. Έχουμε έξι διαφορετικές ρυθμίσεις σε ένα πυλώνα. Μα είναι δυνατόν να μην είναι περίπλοκα τα πράγματα σε έξι διαφορετικές ρυθμίσεις. Τα κράτη-μέλη... Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για κοινή αγροτική πολιτική, να πούμε ότι δεν είναι κοινή αυτή η αγροτική πολιτική αν υπάρχουν τόσε πολλέ διαφορετικέ ρυθμίσει. Δεν έχει τίποτα να κάνει αυτό πλέον με την κοινή αγροτική πολιτική είναι λάθος και η αρχική προσέγγιση. Αν έχουμε να προτείνουμε ένα κατάλογο εκατοντάδων μέτρων, θα πρέπει αυτά τα μέτρα να μπορούν να εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσαρεστημένος που τα ζω αυτά. Εγώ το 2019 δεν θα είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά πώς θα βγουν οι συνάδελφοι να πούν στους αγρότες τι ιδέες αποφασίστηκαν. Και δεν μπορούμε να μιλάμε ότι, και να λέμε ότι έγιναν τα πράγματα απλούστερα. Το Κοινοβούλιο τότε αποφάσισε με 90% ότι δεν θέλουμε ένα νέο σύστημα πληρωμών που θα οδηγήσει σε ένα νέο σύστημα πληρωμών ισχύσεων και κυρώσεων. Και τότε υποστήριξε λοιπόν αυτά ο Επιτροπός Τσιόλος και τελικά έχουμε ένα νέο σύστημα πληρωμών με νέο μηχανισμό κυρώσεων και πληρωμών. Πώς λοιπόν θα βγούμε και θα πούμε ότι μόνο τα γενικές εκτάσεις υποστηρίζονται τελικά τα χρήματα αυτά όμως δεν θα καταλήξουν στον ενεργό αγρότη και αυτή η αγροτική πολιτική λοιπόν θα αποτύχει. Ελπίζω και εύχομαι με τον νέο επίτροπο να ελεγχθούν ήδη από το πρώτο έτος πλήρως να ελεγχθούν αυτά τα κείμενα και να καταλήξουμε σε μια δίκαιη αγροτική πολιτική γιατί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι ανεύθυνο και πολύ λυπάμαι που κι εγώ είμαι συνυπεύθυνος για αυτό το τέρας. Μάλιστα. Ε, μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών έλαβε μέρος σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας των μεταρρυθμίσεων και έχουμε συνέστηση της συνυπευθυνότητάς μας, γιατί είμαστε και εμείς συνδημιουργοί αυτών των μεταρρυθμίσεων. Η κυρία Μαγκίνες. Κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν έλεγα απλώ συμφωνώ με τον Άλμπερντ Ντέσ, δεν θα είχα να προσθέσω τίποτα άλλο. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο τμήμα του προβλήματο, αλλά και τη λύση. Αυτή η λύση, τότε λύση έχει γίνει πρόβλημα για δύο λόγου. Δόθηκε ε, ιδιαίτερη προσοχή στο οικονομικό σκέλος, στον προϋπολογισμό και όχι ε, αρκετή προσοχή στο, στην αντίκτυπο του πρασινίσματος. Εγώ σας προειδοποίησα ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλό για τις ε, περιοχές ε, εστιασμένες ε, στην οικολογία, στο οικολογικό ενδιαφέρον. Και τα μέτρα τελικά δεν είναι φιλικά προς τον αγρότη. Ένας αγρότης ήρθε το Σάββατο στο γραφείο μου και μάλιστα έχει αεροτρές καλλιέργειες μεγάλες και με ένα μονοπάτι δίπλα στο χωράφι του και δίπλα ένα δάσος. Ένα, μια πραγματική ουσιαστικά περιοχή εστιασμένη στην οικολογία. Οι Ιρλανδικές αρχές του είπαν ότι αυτό το μεγάλο τμήμα, ε, παρά το μεγάλο τμήμα του δάσου που είχε δίπλα στην αγροτική του καλλιέργεια, θεωρείται δεν, οι Ιρλανδικές αρχές θεωρούν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για το πρασίνισμα. Θα έπρεπε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση και όχι εστίαση μόνο στο αρωτρέο τμήμα. Και μάλιστα όταν οι τιμές των σιτηρών έχουν πιάσει πάτο, είναι λογικό να είναι δυσαρεστημένοι και να δυσανασχετούν οι γεωργοί. Γιατί τελικά θα οδηγηθούμε σε μη βιώσιμε αγροτικέ πρακτικέ. Θα αναγκάζονται οι αγρότε να έχουν τρει καλλιέργειε αντί για δύο ή μία. Το πρασίνισμα είναι σημαντική καινοτομία, αλλά ο τρόπο που το εφαρμόζουμε οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Γιατί εφαρμόζουμε το πρασίνισμα με λάθο τρόπο. Θα πρέπει η περιβαλλοντική διαχείριση να, γίνει, να αποτελεί τμήμα των ε, βέλτιστων αγροτικών πρακτικών και όχι αυτό που κάναμε. Και αυτό είναι πραγματικά το όνειρο του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να προσλάβουν και άλλο προσωπικό. Αλλά για τους αγρότες που παράγουν το τρόφιμά τους θα είναι εφιάλτης. Νομίζω ότι δεν βρήκαμε τη σωστή ισορροπία. Και επαναλαμβάνω, σας είχα προειδοποιήσει, έπρεπε να καταλήξουμε στη συμφωνία, αλλά εδώ έχουμε δύο εναλλακτικέ. Η μία είναι να ακούσουμε τις εκκλήσεις του Τζιμ Νίκολσον και άλλων, να μην το εφαρμόσουμε από τώρα στους αγρότες, να μην τους τριμώξουμε, για να τους βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό και να αναζητήσουμε το συντομότερο δυνατό αναθεώρηση, σημαντική αναθεώρηση. Θέλουμε φυσικά ε, προστασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορούμε να ενοχλούμε τους αγρότες στις κανονικές τους πρακτικές με μέτρα και μηχανισμούς ελέγχου που τους επιβάλλουμε αδίκως. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή πραγματικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Η κυρία Ντότς, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ μπορώ να πω ότι καταψήφισα την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και εξ αρχής προειδοποίησα ότι είναι υπερβολικά περίπλοκο το σύστημα. Αυτό θα οδηγούσε σε περαιτέρω κυρώσεις και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και ως αποτέλεσμα τα τελευταία τρία σημεία να κοιτάξουμε από την παρουσίαση της Επιτροπής. Λέτε ότι θα δώσετε ενίσχυση και αρρωγή στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ. Πριν από την τρέχουσα εβδομάδα μίλησα με τους υπεύθυνους πληρωμής του τομέα του Υπουργείου Γεωργία στην Ιρλανδία αναμένουν ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές για το πρασίνισμα, για τους ενεργούς ε, γεωργούς, τους νεαρούς γεωργούς και σε ό,τι αφορά θέματα εταιρικής σχέσης. Όλες αυτές οι διευκρινήσεις δεν έχουν καταφτάσει. Παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να εφαρμόσουν όλα αυτά στα κράτη-μέλη και ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Και όπως είπε και η κυρία Μαγκίνες, τελικά αυτό θα οδηγήσει σε κυρώσεις που θα οδηγήσει και με πάσα ειλικρίνεια πρέπει να σας πω ότι η δική μου η περιοχή έχει υποστεί και τέτοιες κυρώσεις τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους που ζήτησαν να καταργηθεί να υπάρξει αναβολή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή γιατί είναι χαοτική η κατάσταση και χαοτική και η έλλειψη πληροφοριών Και όλα αυτά περιπλέκονται περαιτέρω από το γεγονός ότι τελευταία, από ό,τι διαβάζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μέτρα για το τυρί. Είναι εκτός τόπου και χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και μάλιστα τάχιστα για τους γεωργούς, γιατί η κατάσταση πραγματικά είναι εκτός ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γλέζος. Από την ε, εισήγησή σας παρασύρθηκα τόσο πολύ για όσα ωραία είπατε που αφαίρεσα το θα και βρέθηκα σε έναν παράδεισο πράσινο όπου με ξύπνησε ξαφνικά η πραγματικότητα κατάγομαι από ένα νησί των Κυκλάδων, την Άξο, όπου έχει δύο καταπληκτικά προϊόντα. Την πατάτα, είμαστε παραγωγή πατάτας και σπόρου πατάτας και του περίφημου κίτρου που δεν υπάρχει ως εσπεριδοειδές σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αλλά ξαφνικά μας είπανε ότι ένα καινούριο φυτό σας δίνουμε για να καλλιεργήσετε και ποιο είναι αυτό το καινούργιο φυτό, είναι τα φωτοβολταϊκά της Μέρκελ επειδή θέλει να πάρει από την Ελλάδα ηλεκτρισμό γιατί η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια από όλες τις χώρες της Ευρώπης τη μεγαλύτερη. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση γιατί πολλές φορές θα ερωτήματα και απάντηση δεν πήρα. Πώς θα ξεφυτρώσουμε τα φωτοβολταϊκά που καλύπτουν τα πατατοχώραφα και θα ξαναγυρίσει η γη στον προορισμό της να καλλιεργεί την πατάτα και το κίτρο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ. Μία μικρή παρατήρηση για μας. Είμαστε μέλη της Επιτροπής και θα έπρεπε να μην ξεχνάμε με όλη την κριτική που κάνουμε ότι είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι για τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε υπόψη. Ακούσαμε ότι αν πρέπει να πούμε στους αγρότες τι προέκυψε από την, τελευταία, από την τελευταία μεταρρύθμιση, τελικά τι προέκυψε, λίγο λιγότερα χρήματα, λίγο περισσότερη γραφειοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί το στόχο μας για την ε, πολιτική. Γιατί τελικά δεν θα έχουμε καθόλου χρήματα στο τέλος και μόνο γραφειοκρατία. Ρωτώ λοιπόν, γιατί εγώ έλεγα ε, από την αρχή ότι δεν πρέπει να μπει το greening αυτό το πρασίνισμα στην πρώτη πυλώνα. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ενδιαφέρει αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση πραγματικά, όπου θα ήσασταν αντιτεθειμένοι να βρείτε τα σφάλματα και να παραδεχτούμε ότι επιβαρύναμε τον πρώτο πυλώνα με πράγματα που δεν ανήκαν σε αυτόν και σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι πήγαν λάθος τα πράγματα αυτά, να διορθώσουμε τις εσφαρμένες αποφάσεις που ελευθύσαν. Σας ευχαριστώ. Ωραία το διατυπώσατε ότι επιβαρύναμε υπερβολικά τον πρώτο πυλώνα. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη αυτή η κρίση. Ο κύριος Άντριου. Oui, merci, euh, président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ την κριτική την οποία ασκούμε στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Έχουμε πράγματι εργαστεί πάνω στο αρχικό κείμενο που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως ακούστηκε στα πλαίσια της παρουσίασης βρισκόμαστε σε φάση συναπόφασης μέσω του τριμερούς διαλόγου και δεν μπορούμε εμείς να αγνοήσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Κατανοώ και την περιπλοκότητά τους αν θέλετε, αλλά αυτό το οποίο με λυπεί βαθύτατα είναι ότι πέρα από τα πολιτικά κείμενα πάνω στα οποία συμφωνήσαμε ή μη με το Συμβούλιο, η μετατροπή τους σε πρακτικές ρυθμίσεις που έγινε είναι η επόμενη πράξη αν θέλετε που έχει άμεση σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις Και εδώ βλέπουμε ότι η μετάβαση, η, δεν υπάρχει ταύτιση ή δεν υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα σε αυτά που είχαμε ψηφίσει και στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Καταρχάς, παράδειγμα, αδειοδοτήσεις για τα αμπελοϊνικά. Ε, δεν καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και δεύτερο θέμα αφορά τους μόνιμους βοσκοτόπους, αλλά όπου δεν κυριαρχεί ακριβώς ε, ένα είδος ε, καλλιέργειας. τι εννοώ με αυτό. Έχει υπάρξει μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου υπήρξαν συζητήσεις για τις μη κυρίαρχα χορτολιβαδικές τέτοιου είδους εκτάσεις και στο κείμενο του Καπούλα Σάντος και στα πλαίσια του Συμβουλίου ε, του 12. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για τον νότο της χώρας μου και τις μεσογειακές περιοχές. Και από ό,τι φαίνεται ε, δεν θα είναι επιλέξιμες πλέον οι εκτάσεις αυτές αυτό σημαίνει ότι η πολιτική και η οικονομική ανάλυση που είχαμε κάνει στα εδάφια αυτά, για τα εδάφια αυτά, και εδώ θα συμφωνήσουν και οι Σκότοι και, και ίσως και κάποιοι άλλοι, Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές όπου κυριαρχούν οι βελανιδιές ή κυριαρχούν οι καστανιές θα θεωρούνται χορτολιβαδικές οι εκτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σανέλ. Σανίλ. Σανίλ. Σανίλ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, μια και είμαι νέο ε, βουλευτή εδώ στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα λοιπόν να πω εξ αρχή το εξή, ότι γνωρίζω πολλού εδώ στην αίθουσα, αλλά εγώ δεν συμμετείχα σε αυτά που αποφασίστηκαν και συζητήθηκαν τα τελευταία 10-12 χρόνια. Στο Υπουργείο Γεωργίας στην Ουγγαρία, πριν από 10-12 χρόνια γνώρισα καλά το σύστημα αυτών των άμεσων ενισχύσεων. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Τελικάστρο και θα πρέπει να το δούμε αυτό σε ιστορικό πλαίσιο. Εξ όσων θυμάμαι, τότε η κοινή αγροτική πολιτική είχε θέσει δύο στόχους βασικούς. Καταρχάς, να διασφαλίσουμε την επιβίωση του αγρότη και μία σίγουρη παραγωγή και κατά δεύτερον ο λαός, οι λαοί της Ευρώπης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευνοϊκές ε, τιμές και σε ποιοτικά προϊόντα. Αυτοί ήταν οι δύο στόχοι, οι οποίοι εντωμεταξύ έχουν διαχωριστεί ο ένας από τον άλλον και μέσω των άμεσων ενισχύσεων μπορέσαμε με να πετύχουμε μια κάποια μακροπρόθεσμη ασφάλεια για τους αγρότες. Ξέρω ότι υπάρχουν και αγρότες που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά συνολικά θα έλεγα ότι είχαν καλό αντίκτυπο σχετικά αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές και Πρέπει να πω αφετέρου ότι στην Ευρώπη βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος πεινάει, υποσυτίζεται, ζει σε καθεστώς στόχιας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις αιτιώδεις συνάφειες. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει ιδιαίτερος και το οποίο θα ήθελα εδώ και πολύ καιρό ήθελα να θέσω στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όταν βλέπει ο πολίτης ως καταναλωτής τι συμβαίνει εδώ, έχει νόημα από τη μία να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για άμεσες ενισχύσεις, δισεκατομμύρια. Και από την άλλη να φορολογούμε τόσο έντονα και τόσο, με τόσο υψηλού συντελεστέ τα τρόφιμα. Υπάρχουν χώρες όπου είναι μηδενικός ο συντελεστής του ΦΠΑ, αλλά στη χώρα μου πληρώνουμε 27% ΦΠΑ για τα τρόφιμα. Και μεταξύ των δύο αυτών άκρων, μεταξύ του 0% και του 27% υπάρχουν ασφαλώς και πάρα πολλές ενδιάμεσες λύσεις. Θα έπρεπε λοιπόν οι γεωργοί να ενισχύονται από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη ο φόρος προστατεύμενης αξίας για το τρόφιμα είναι πολύ διαφορετικός στις χώρες της Ευρώπης. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρόφιμα είναι κάτι παρόμοιο όπως τα φάρμακα. Ε, χρειάζονται στο σώμα μας πολύ απλά. Και θα μπορούσαμε ίσως σε κάποιο βαθμό έτσι να περιορίσουμε τα κράτη-μέλη και να εισαγάγουμε ένα ανώτατο συντελεστή φορολόγηση των τροφίμων. Και έτσι λοιπόν θα ήταν πιο εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Σράιερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, μιλάμε για την υποστήριξη των αγροτών, αλλά θεωρώ ότι το θέμα είναι και η υποστήριξη της πολιτικής. οδεύουμε στο 2020. Όταν μιλάμε για γόρδιωτισμούς και για την επίλυσή τους, δεν θα έπρεπε στην Ευρώπη να κοιτάξουμε πώς ε, επιβάλαμε τις ε, περιφέρειες Natura 2000, για παράδειγμα, συγκεκριμένες περιοχές. Νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να οδεύσουμε. Και κάτι άλλο που ισχύει για την περίοδο της κρίσης. Πρέπει να σας πω ότι στην Ολλανδία συναντιέμαι με πάρα πολλούς ε, που είναι επιχειρηματίες που δεν ήξεραν ποτέ ότι είχαν δικαίωμα να έχουν τέτοιες ενισχύσεις. Θα έπρεπε δηλαδή να εξηγήσουμε πολύ πιο καλά τι υποστηρίζουμε. Υποστηρίζω την ευρωπαϊκή πολιτική, υποστηρίζω την ΚΑΠ, αλλά όταν μιλάμε για πολίτες πρέπει να έχουμε υπόψη και την κριτική που ασκούν. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε όλα αυτά απεικοδομητικά. Καταλαβαίνω τι λέει ο Άλμπερτες και συμφωνώ ότι είναι γραφοκρατικό το έκτρομο αυτά. Αλλά κοιτάξτε, ε, έχω και εγώ γνωρίζω κόσμο που έχει λογιστές και τα βγάζουν άκρη με αυτά τα γραφειοκρατικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση αυτή. Πολλά ακούσαμε από διάφορους συναδέλφου. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με πολλού εξ αυτών, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή ε, και να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ε, ήθελα να ξέρω πώς τα διάφορα κράτη-μέλη θα εισαγάγουν τα μέτρα πρασινίσματος, γιατί έχω την αίσθηση και πολύ ανησυχώ ότι θα εισαχθεί με διαφορετικό τρόπο. Και πώς θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και να παραμείνουν ίσοι οι όροι του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και θέματα τοπίου σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα έχει να κάνει αυτό δηλαδή με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες με τις οποίες δεν έχουν καν διάθεση να ασχοληθούν οι θύνοντες από τα Υπουργεία. Συγκεκριμένα λοιπόν τι γίνεται με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κατά δεύτερον, όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, μπορούμε να πούμε ότι το 2015 μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει αυτή η περίοδος του πρασινίσματος. Είναι αυτό υπεύθυνο. Οι αγρότες προσπαθούν να σχεδιάσουν τις επόμενες οδιές τους. Δεν ξέρω όμως κανέναν αγρότη που τελικά να γνωρίζει πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το πρασίνισμα, μήπως τα Υπουργεία, μήπως εσείς ξέρετε πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η κατάσταση. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, τουλάχιστον στη δική μας χώρα. Υπάρχουν διάφορα γραφεία συμβουλευτική που θα βγάλουν χοντρά λεφτά από τους αγρότες. Γιατί οι αγρότες θέλουν να ξέρουν τι θα κάνουν και τι πρέπει να κάνουν. Και θεωρώ ότι αυτό είναι παράδεκτο. Κατά δεύτερον, αναφερθήκατε σε αυτόν. Ένας ε, αγρότης ε, που θέλει να ρυθμίσει τα πράγματα στη δουλειά του καλά. Προσπαθεί να εφαρμόσει τα μέτρα πρασινίσματος και μετά εκ των υστέρων όντω μπορεί να κρυθεί από το εθνικό συνέδριο ότι δεν το έκανε καλά τα πράγματα και τελικά να υποστεί τι συνέπειε. Α μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πώ μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Και τελευταία ερώτηση, συμφωνώ με την ερώτηση του Πέτερ Γιάρ. Να αξιολογήσουμε τι γίνεται και σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι αυτά τα στοιχεία πρασινίσματος ταιριάζουν πιο καλά στο δεύτερο πυλώνα, εκεί να μπουν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ είμαι καινούριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δέκα όμως χρόνια εργαζόμουν στον Εθνικό Οργανισμό Ελέγχου. Και μάλιστα προ... ήμουν και πρόεδρος τοπικού συμβουλίου και οργάνωσα πολλά σεμινάρια για την εφαρμογή των κανόνων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Γι' αυτό ξέρω και τα υπέρ και τα κατά της. Είναι σημαντικό πάντως να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κοινή αγροτική πολιτική, γιατί θέλουμε μια πολιτική που θα λειτουργεί εύρυθμα, που δεν θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και θα πρέπει να διατρανώσουμε τους στόχους μας. Τι θέλουμε να πετύχουμε με το νέο σύστημα και θα τα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους νέους μας στόχους. Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί συνήθως οι αγρότες καλλιεργούν προϊόντα, φυτίες που είναι και πιο προσοδοφόρες, που θα τους αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος. Θα πρέπει να φροντίσουμε όμως για, για την αποζημίωση των ζημιών τους. Γιατί σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις καθυστερημένες πληρωμές και για το πόσο δυναπαθούν οι αγρότες εξαιτία της καθυστέρησης στις πληρωμές. Οι αγρότες θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τι γίνεται όταν ξεσπάει μια κρίση. Για παράδειγμα το ρωσικό εμπάργκο. Με το νέο σύστημα θα διευκολυνθεί η κατάσταση για τους αγρότες θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών μας και ίσες συνθήκε ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρτέ. Σα uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Δεν ξέρω αν αυτό το PowerPoint, η παρουσίαση αυτή μας έχει αποσταλεί. Ίσως θα μπορούσε να γίνει έστω και μετά από τη συνάντηση. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκράτησε τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει ένας πολύ ψηλό κίνδυνος κάποια θετικά στοιχεία της κοινή αγροτικής πολιτικής να σκιαστούν από τις αρνητικές εμπειρίες τις οποίες καλούνται να βιώσουν οι γεωργοί. Ε, οι προτάσεις οι οποίες που έγιναν για πιθανή αναβολή του greening είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό και το τι μπορεί να ακολουθήσει ως προς το λεγόμενο greening. Όλοι έχουν αρχίσει να σκέπτονται και την πιθανή, ε, ε, τον πιθανό έλεγχο και την αξιολόγηση που θα πρέπει να γίνει. Αυτό θα οδηγήσει σε μια πλήρη νέα μορφή ελέγχου των πολιτικών ή θα είναι κάτι το τυπικό. Θα υπάρξει επιτέλους η απαιτούμενη προσοχή για τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Θυμίζω ότι ιδιαίτερα στην ΚΑΠ κάθε δύο χρόνια όλοι λένε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο γραφειοκρατίας, το οποίο έχουμε ρίξει πάνω στις πλάτες των γεωργών και υπάρχουν πάρα πολλοί μικροί γεωργοί σε επίπεδο ε, γραφειοκρατίας ε, καλούνται να κάνουν τεράστια, τεράστιες προσπάθειες συμπλήρωσης ε, εγγράφων, τεκμηριώσεων και τα λοιπά αντίστοιχες των μεγάλων βιομηχανιών. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν πρέπει να μην αγνοήσουμε, είναι μια φεά περιοχή για όλους, είναι οι ευθύνε ε, ε, της Επιτροπής και της κοινότητας και το είπε και η Μαγκίνας. Εγώ είμαι υπέρ της εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με ξεκάθαρο τρόπο και προς τους ε, υπευθύνου σε κάθε χώρα αλλά και προς τους ίδιους τους γεωργούς να γνωρίζουν το ποιος είναι υπεύθυνο και σε ποιο επίπεδο γιατί. Ε, δεν ε, περιόρισα τους ομιλητές ε, και βρίσκομαι τώρα σε δύσκολη κατάσταση, σε δύσκολη θέση. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε αυτά που ακούσαμε και ιδιαίτερα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες επικρίσεις συνέχεια. Γιατί αρκεί μία φορά η Κομισιόν τα σημειώνει όλα αυτά. Ο κύριος Λουαζό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εμπαρόδο να διευκρινίσω ότι είμαι και εγώ Γάλλος γεωργός και με επηρεάζει αυτή η αγροτική πολιτική. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Γαλλίας, στη μεγαλύτερη σιτοπαραγωγό περιοχή της Ευρώπης. Και έχω σοβαρούς λόγους ανησυχίας. Μιλούμε για ένα νέο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων. Μα τι μου λέτε. Ε, και ταυτόχρονα ενισχύουμε την αιρεσιμότητα με βάση το περιβάλλον, της εκμεταλλεύσιμες καλλιέργειες. Έξι καθεστώτα, τρία προαιρετικά, τρία υποχρεωτικά. Κατάργηση των ποσοστώσεων. Εντάξει, δεν είναι καινούριο, αλλά η κατάργηση των γαλακτοκαμπικών ποσοστώσεων είναι χρονικό ανακερθούντος θανάτων των γαλακτοπαραγωγών. Όλα αυτά είναι μορφές απολυταρχισμού, ολοκληρωτισμού. Αποτέλεσμα περισσότερη γραφειοκρατία, περιορισμοί, περισσότερη έλεγχη και σας ερωτώ. Πού βρίσκεται η γραφειοκρατική απλούστευση που μας υποσχεθήκατε. Όλο γι' αυτό ακούμε, αλλά δεν τη βλέπουμε. Κάθε χρόνο, εδώ και 22 χρόνια, η Γαλλία δίνει 20, 20 δισεκατομμύρια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 13 δισεκατομμύρια πάνε στη Γεωργία. Υπάρχει όμως μια διαφορά 18 δισεκατομμύριων εδώ. Πόσο καιρό θα πληρώνει τους λογαριασμούς η Γαλλία, για πόσο καιρό ακόμη. Ενώ ταυτόχρονα οι ενισχύσει μειώνονται. Οι τιμές πέφτουν. Για να μην μιλήσουμε για το ρωσικό εμπάργο που επιδεινώνει την ήδη ολέθρια κατάσταση. Πώς θα μας προστατεύσει όλα αυτά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού μας προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού φροντίζει για τους α, Γάλλους γεωργούς. Είστε ανεύθυνοι. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι για πόσο καιρό ακόμη οι Γάλλοι γεωργοί θα είναι οι θυλάζουσες, οι γαλακτοφόρες αγελάδες μάλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής προς Θεού. Ε, μιλήσατε για τους ε, Γάλλους Γεωργούς. Ε, νομίζω είναι υπερβολικά αυτά που είπατε, για να το πω κατεφημισμόν υπερβολικά. Στην κοινή αγροτική πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι επωφελούνται. Αυτό φαίνεται από επιστημονικές μελέτες. Παρακαλώ λοιπόν λίγο, λίγη αντικειμενικότητα. Ας μην κάνουμε επικρίσεις ε, ε, ο ένας μετά τον άλλον. Συμφωνήσαμε να καταργηθούν οι ποσοστώσεις, ε, να καταργηθούν κάποια ανώτατα όρια, κάποιες ενισχύσεις. Παρακαλώ, λίγη αντικειμενικότητα. Λυπούμε που παρενέβηνε εδώ, αλλά και εγώ παρακολουθώ την Ευρωπαϊκή Γεωργία 10 χρόνια. Παρακαλώ, ας είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι νέα Ευρωβουλευτής από την Κροατία και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη θέση των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Βλέπω στις μεταρρυθμίσεις για την κοινή αγροτική πολιτική ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις δεν λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Ερωτώ λοιπόν τι γίνεται με αυτή την προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας εις βάρος όμως της ιδιαιτερότητας και της ποιότητας. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες στις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τους ε, αγρότες ή τους ανθρώπους που μένουν στα χωριά άσχετα με την ηλικία τους, γιατί μερικοί άνθρωποι θυσίασαν όλη τους τη ζωή στη γεωργία και στη γεωργική παραγωγή και είναι κρίμα να περιθωριοποιούνται στην κοινή γεωργική, από, την κοινή αγροτική πολιτική εφόσον δεν είναι πια ενεργοί γεωργοί και εφόσον πια ασχολούνται με κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που μένουν στην Ήπεθρο, στα χωριά, πρέπει να τύχουν υποστήριξη, ακριβώς επειδή ζουν εκεί. Και διαφυλάσσουν το χώρο, διαφυλάσσουν τα χωριά, την Ήπεθρο, διαφυλάσσουν την βιοπικιλότητα, τη ζωή, την ποιότητα των τροφίμων. Αυτά θα πρέπει να τα εκτιμήσουμε και να τα επιβαραβεύσουμε. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα χωριά μας να ερημώνονται και τα μόνα τρόφιμα να τα λαμβάνουμε από τη βιομηχανική παραγωγή και όχι από τους γεωργούς μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράντ. Oui, monsieur le president euh, Ναι, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω κάποια βασικά πράγματα. Η Γαλλία όχι μόνο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης εξ αρχής, αλλά είναι η πρώτη γεωργική χώρα της Γαλλίας και είναι η δεύτερη συνεισφορέα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάτε για τη Γαλλία να προσέχετε, γιατί οι γεωργοί της Γαλλίας φύγονται περισσότερο από ίσως άλλους. Λοιπόν, να προσέχετε. Δεύτερον τώρα, σχετικά με την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα μετά από αυτά τα οποία είπατε, οι γεωργοί κατάλαβαν ότι τα προβλήματά τους τελικά τα δημιουργεί εν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό στις εκλογές θα σας ε, περπιθούν ανάλογα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με τον νέο Επίτροπο. Όλα γίνονται για να συστηματοποιήσουμε τη λογική της υπερφιλελεύθερης αγοράς. Είδαμε τι έγινε με τις ποσοστώσεις. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όλα αυτά που είπατε είναι εις βάρος των γεωργών. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το νέο Αμερικανικό νόμο για τη γεωργία, το νέο Farm Bill, από συνδεδεμένες πληρωμές και θα παράγουν χάνοντας χρήματα σε περίπτωση κρίσης γιατί δεν θα υπάρχει ελάχιστη τιμή. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση τίποτα δεν θα μπορεί να γίνει. Αν ψάχνετε για λύση λοιπόν και αν δεν έχετε ιδέες, αυτό που έχω να σας πω κύριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι σήμερα τα κράτη θα πρέπει να ανακαλύψουν τις στρατηγικές τους και να ρυθμίσουν τις χρηματαγορές βοηθώντας τις παραγωγές τους, μόνες τους οι χώρες. Συμφωνώ με το δεύτερο τμήμα της παρέμβασής σας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Ο κύριος Χόισλινγκ. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κάποιε προσωπικέ παρατηρήσει. Με ε, ενοχλεί το γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ενεργοτική μεταρρύθμιση γιατί συγκεντρώθηκε τελικά πλειοψηφία και από το ΕΛΚ και από του σοσιαλιστέ στο Κοινοβούλιο υπέρ της μεταρρυθμίσης. Και ε, τώρα όλοι αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα να κάνουν. Δεν είναι δυνατόν να αναλαμβάνουμε έτσι πολιτική ευθύνη. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα σήμερα. Και αυτό οφείλεται, κυρίε και κύριοι, στο γεγονός ότι κάναμε και εκατοντάδες τροπολογίες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα δηλαδή να κατηγορούμε τον Επίτροπο μόνο, νομίζω ότι είναι κάπως απλοϊκό. Φυσικά, αν ε, ρωτήσουμε τους γεωργούς αν είναι τα πράγματα πολύ περίπλοκα, τι θα ήθελα να... Ε, οι γεωργοί να του δίνουμε τα χρήματα στην αρχή χωρίς να υπάρχει έλεγχος αλλά ειλικρινά επρόκειτο ποτέ να λειτουργήσει τέτοιο σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε και ένα σύστημα ελέγχου. Χρειάζεται και κάποια αντιστάθμιση. Αυτό ήταν από την αρχή η συμφωνία. Δεν θέλω να κατηγορήσω τόσο πολύ τον Επίτροπο όπως ο Άλμπερντες, γιατί με πάσα ειλικρινή να πούμε ότι για να, να δεν μπορούσε να διατηρηθεί στο επίπεδο που ήταν ο αγροτικός προπολογισμό. Εμείς όλοι μαζί τα πετύχαμε σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των αξιώσεων. Φυσικά λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον πώς θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε που θα αφαιρέσουν την εξάρτηση των γεωργών από τον πρώτο Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν τα ταμεία στη τελική ανάλυση. Κανένα άλλο κλάτος δεν υποστηρίζεται τόσο πολύ από άμεσες ενισχύσεις. Όλοι όσοι λοιπόν κατηγορούν αυτή τη μεταρρύθμιση να το σκεφτούν δύο φορές, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, νομίζω ότι λασπολογούν κατά της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Πολύ ε, βαθιστόχαστα και ισορροπημένα τα σχόλια. Κυρία Μόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα ένα πολύ μεγάλο του τμήματος των ενισχύσεων προς τους γεωργούς στην πατρίδα μου και ιδιαίτερα στη Σαρδινία δημιούργησε στη γέννηση μιας μεγάλης σειράς από απάτες, από κομπίνες. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν χιλιόμετρα νομοθετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μια υποχρεωτική και μόνιμη προσφυγή σε εμπειρογνώμονες, σε συμβούλους, οι οποίοι και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο βρήκανε ε, την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά εις βάρος των γεωργών οι οποίοι έχουν πάντα ανάγκες όλο και μεγαλύτερες. Με αυτό το νέο σύστημα λοιπόν των άμεσων ενισχύσεων θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις απάντες. Έχετε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο, έχετε κάτι σκεφτεί για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουντάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός και δεν θα πω όπως ο Σολομώντας, ο βασιλιάς Σολομώντας, ότι όλοι έχουν δίκιο. Οι συζητήσεις αυτές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ χρήσιμες γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους ψηφοφόρους μας, ε, μεταξύ άλλων και τους γεωργούς μας και όταν έρχονται και μας ρωτάνε θα πρέπει να τους δώσουμε μία απάντηση. Μας ρωτά συχνά για τα μέτρα αυτά του πρασινίσματος. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πολύ πυκνή και περίπλοκη. Και εγώ τα έχω χαμένα μερικές φορές ε, και δεν μπορώ να βρω τον μπούσουλα μέσα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι περίπλοκη κατάσταση και μερικές φορές ε, οι γεωργοί κινδυνεύουν να πληρώσουν πρόστιμα πολύ ψηλότερα από τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Όπως είπε και η κυρία Μαγκίνες, είμαστε και εμείς τιμά της λύσης ε, με τα μέτρα που προτείνουμε. Σίγουρα το 2012 και το 2013 έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, της αγροτικής πολιτικής μας. Αλλά Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των χωρών μελών, ιδιαίτερα μεταξύ δυτικών και ανατολικών, για τις άμεσες ενισχύσεις. Όλοι παραπονιούνται για τα χρήματα, για τις πληρωμές, όλοι διεκδικούν υψηλότερες ενισχύσεις και εκεί υπάρχει ένα κενό. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιταχύνει την διαδικασία ενοποίησης του συστήματος για να έχουμε ομοιόμορφο διαδικασία πληρωμών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς ε, θα δημιουργηθούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, κάτι που είναι απευκταίο. Ευχαριστώ, κύριο Άγνιου. Ευχαριστώ. Αναμασάμε, κύριε Πρόεδρε, τις συζητήσεις για τα καλά της κοινή αγροτικής πολιτικής. Να πω σε αυτούς που ήταν εδώ την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, πως είχα καταθέσει 10 τροπολογίες για την κατάργηση, την απαγόρευση των κατεξουσιοδότηση πράξεων και κανένας δεν τις υποστήριξε τις τροπολογίες αυτές και τώρα γκρινιάζεται. Λοιπόν, άκουσα και έναν Έλληνα βουλευτή που έλεγε ότι στην Ελλάδα του ζητούν να, να αντικαταστήσουν τις καλλιέργειές τους με τα φωτοβολταϊκά και για σε εμά το κάνουν αυτό. Διαρωτώ με λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικές φορές αυτές οι μονάδες παραγωγής είναι γύρω στα 100 εκτάρια. Τι γίνεται ε, ε, για το έδαφος το, πάνω στο οποίο έχουν σε εισαγωγικά φυτέψει. Είναι επιλέξιμες οι περιοχές αυτές ή δεν είναι. Δεύτερον, άκουσα επίσης τον Ούγκρο Ευρωβουλευτή εκ δεξιών, ο οποίος είπε ότι στην χώρα του υπάρχει 27% ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ο κόσμος πεινά σε κάποιες περιοχές της χώρας και αναρωτιέμαι πώς γίνεται κάτι τέτοιο. Όταν ξαφνικά οι κυβερνήσεις σας βάζουν τέτοιου είδους ε, επίπεδα αφορολόγηση ε, είναι προφανές ότι δεν μπορούν ποτέ να τα καταργήσουν. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μπογκόβιτς είναι ο τελευταίος ομιλητής σε αυτό το γύρο των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επενέσω αυτή τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και κυρίως ε, τα μέτρα για την ενίσχυση των νέων, των νεαρών γεωργών. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα για το μέλλον. Και γι' αυτό είμαι υπέρ των μεταρρυθμίσεων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εμείς στη Σλοβενία έχουμε σχεδόν 900 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο σε ό,τι αφορά την αναλογία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και η οικολογο, οικολογικοποίηση αυτών των εδαφών που είναι περιορισμένα και στη Σλοβενία. Αναφέρθηκαν οι, μόνιμες, οι μόνιμοι βοσκότοποι και λιμόνες, ίσως τα μέτρα αυτά δημιουργήσουν κάποια προβλήματα στην εφαρμογή τους. Προβλήματα όμως υπάρχουν και στη διοίκηση. Και αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν τους γεωργούς μας που υποβάλλουν αιτήσει για πληρωμή, αλλά απορρίπτονται επειδή δεν ακολούθησαν όλες τις διατυπώσεις σωστά. Είναι μεγάλη η γραφειοκρατική επιβάρηση για τους αγρότες μας. Οπότε, κατά τη λήψη των νέων μέτρων, παρακαλώ φροντίστε ώστε η διαδικασία να είναι όσο πιο απλή γίνεται. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το γύρο των ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις άμεσες ενισχύσεις και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια σύντομη απάντηση. Δεν έχουμε χρόνο για διεξοδικές απαντήσεις, φαντάζομαι θα τις λάβουμε αργότερα αυτές. Ευελπιστώ πάντως ότι στις, για τις επόμενες παρουσιάσεις δεν θα υποβληθούν τόσο πολλές ερωτήσεις και θα έχουμε χρόνο για πιο διεξοδικές απαντήσεις. Παρακαλώ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος στις απαντήσεις μου. Θα προσπαθήσω να σταθώ στις βασικές ερωτήσεις οι οποίες έχουν επανειλημμένα τεθεί. Σας ευχαριστώ καταρχάς για τις ερωτήσεις σας γιατί δείχνει το τεράστιο ενδιαφέρον που έχετε για το συγκεκριμένο θέμα και για το νέο σύστημα των άμεσων ενισχύσεων που θα τεθεί σε ισχύ από το 2015. Το πρώτο θέμα το οποίο απασχόλησε πολλούς από τους ε, παρεμβαίνοντες έχει σχέση με την ανάγκη απλούστευσης της πολιτικής αυτής. Συνειδητοποιούμε πλήρως αγαπητοί κύριοι τις δυσκολίες οι οποίες έχουν εκφραστεί από πλευρά σας σχετικά με τον αποτελεσματικό τρόπο ε, εφαρμογής αυτής της νέας πολιτικής. Έγιναν κάποια θετικά βήματα για τους μικρούς γεωργούς, για την αιρεσιμότητα. Αλλά θα πρέπει να παραδεχτώ πρώτος ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή και ιδιαίτερα με το λεγόμενο greening στον πρώτο πυλώνα, όπως αποφασίστηκε από τους συνομοθέτες, είναι σαφές ότι για μας και για σας και για όλα τα κράτη-μέλη είναι μια δύσκολη υπόθεση. Στην παρούσα φάση λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ και αρκετούς μήνες για να τα θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή. Να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω εδώ λίγο το σε, σε τι οφείλεται αυτή η περιπλοκότητα. Βρισκόμαστε σε ένα διακανονιστικό πλαίσιο πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι στο παρελθόν. Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική πιο αποδοτική, πιο στοχευμένη, πιο πράσινη, που να ανταποκρίνεται πολύ πιο άμεσα σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ως εκ τούτου πρέπει να λάβουμε ακριβώς τις δυνατότητες της τοπικές υπόψη. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν για πρασίνισμα, Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία προς τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τώρα σε μια Ευρώπη των 28, να ανταποκριθούμε λοιπόν καλύτερα στις ανάγκες των περιοχών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Υπέθρου. Όποιος θέλει πιο σωστή ε, πολιτική, πιο σωστή στόχευση και μεγαλύτερο πρασίνισμα, αυτό σημαίνει και μεγαλύτερες περιπλοκές στους ελέγχους τουλάχιστον. Και εδώ συνεργαζόμαστε και μαζί σας και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να βρούμε την πιο σωστή ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις της συγκεκριμένης αυτής πολιτικής, στην επίτευξη των στόχων αυτής της νέας πολιτικής, με μια ε, υγιή δημοσιονομική διαχείριση, γιατί να μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για πολύ υψηλές πιστώσεις. Και αυτό δημιουργεί επιπτώσεις γραφειοκρατικές και για τις εθνικές διοικήσεις και φυσικά για τους ίδιους τους γεωργούς. Προσπαθούμε λοιπόν να εργαστούμε στενά με το σύνολο των κρατών μελών, μέσω workshops, μέσω διασκέψεων, μέσω διμερών επαφών, μέσω απαντήσεων σε ερωτήσεις που μας τίθενται. Συνεργαζόμαστε με τις περιφερειακές επίσης αρχές για να εφαρμόσουμε με σωστό τρόπο αυτή τη νέα πολιτική και αυτό το νέο σύστημα πρασινίσματος και αν πάρω το παράδειγμα της Ιρλανδίας ε, και της, της ε, Δημοκρατίας αλλά και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι μια χώρα την οποία επισκεφθήκαμε δύο φορές, είναι μια χώρα την οποία θα επισκεφτούμε για τρίτη φορά για να βοηθήσουμε τις εθνικές και τις τοπικές αρχές και τις περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν σωστά το νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων. Αύριο ξεκινάει ένα, μια στρογγύλη τράπεζα η οποία θα κρατήσει 10 μέρες σχεδόν για την σωστή εφαρμογή και ερμηνεία του νέου ολοκληρωμένου συστήματος, του ΙΑΚΣ, στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς μας. Στο εσωτερικό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας δημιουργήθηκε μια νέα υπηρεσία στήριξης των κρατών μελών, οι προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά είναι σημαντικό μετά από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, μετά από την πρώτη αξιολόγηση τέλος 15 αρχές 16, να προσπαθήσουμε να δούμε με πιο πρακτικό τρόπο, με πιο λειτουργικό τρόπο τέθηκε σε λειτουργία η πολιτική αυτή και ανάλογα με τις ανάγκες να δούμε τι στοιχεία θα πρέπει να διορθώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε ε, αντίθετα λοιπόν με αυτά τα οποία ακούστηκαν, με κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν, αυτή η αξιολόγηση του greening σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα είναι μια αναθεώρηση, μια εξέταση πολύ σοβαρή από πλευράς των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα τρίτο στοιχείο πάνω στο οποίο θέλω να σταθώ αφορά τις διάφορες ε, αναφορές που έγιναν σχετικά με την αναβολή της εκκίνησης της διαδικασίας greening για το 2016. Είναι σαφές πως την παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο, βλέποντας το ισχύον διακανονιστικό πλαίσιο, να μην πω ανέφικτο, να αναβάλει κανείς για ένα χρόνο το greening αλλά να θυμίσω επίσης που υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές ρυθμίσεις και με το EX και με το σύστημα ελέγχου που προβλέπουν μια σταδιακή εφαρμογή του συστήματος τα επόμενα τρία χρόνια. Προβλέπεται ήδη δηλαδή η διαδικασία του greening να μην καταστεί ε, λειτουργική κατά 100% παρά μόνον από το 2018 Υπάρχει δηλαδή μια μεταβατική προβληπόμενη περίοδος. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα λοιπόν της αναβολής της εφαρμογής της διαδικασίας σε εισαγωγικά πρασινίσματος. Τώρα για την υποστήριξη στην οικογενειακή γεωργία, για την υποστήριξη στους νέους γεωργούς, ε, για την υποστήριξη των μεσογειακών περιοχών οι οποίες δεν βασίζονται αποκλειστικά σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Νομίζω ότι εμείς αναγνωρίζουμε πλέον ότι η οικογενειακή γεωργία είναι η βάση της γεωργικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και η ευρωπαϊκή πολιτική ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων γεωργών και με τον πρώτο και με το δεύτερο πυλώνα για τις μόνιμες εκτάσεις αυτές στις μεσογειακές περιοχές όπου βλέπουμε αρκετές περιοχές που δεν είναι καλυμμένες από χόρτο Νομίζω ότι εδώ οι εφαρμοστικές πράξεις και η κατεξουσιοδότηση πράξεις μπορεί να διορθώσουν ότι δεν πάει καλά. Θα σταματήσω εδώ Πρόεδρε. Αυτά ήταν τα βασικά τα οποία τέθηκαν για το δικό μου κομμάτι. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση. Την παρουσίαση του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς. Θα μας κάνει την παρουσίαση ο Διευθυντής Χέρμαν Φερστέινεν. Παρακαλώ, μην ξεπεράσετε το δεκάλεπτο. Και μετά η ερωτήση θα είναι ενός λεπτού. Ελπίζω να προλάβουμε. Και μάλιστα θα είναι και καλή εξάσκηση για μας πριν από την ακρόαση. θα μιλάμε, λίγο θα ακούμε και έτσι θα προετοιμαστούμε καλά και για την ακρόαση. Εν είναι έτοιμος ο Διευθυντής, του δίνω το λόγο για την παρουσίαση. Θα ζητούσα πάντως περισσότερη πειθαρχία σε αυτό το δεύτερο γύρο, στη mm. δεύτερη παρουσίαση. Κύριε Φερστέιλεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση και γρήγορη του θέματος. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικές διαφάνειες που είναι σημαντικές για να δούμε τις αγορές και την ανταγωνιστική μας θέση. Τι καταφέραμε μετά από 30 χρόνια μεταρρυθμίσεων. Ξεκινώ με την διαφάνεια για τις τιμές αραβώσιτου και σιτού βλέπετε τις τιμές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη σύγκληση των τιμών, κάτι που σημαίνει ότι η δική μας ε, τιμή για το ΣΥΤΟ είναι παρόμοια με την παγκόσμια τιμή ΣΥΤΟ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για τους ε, κτηνοτρόφους μας, ώστε να έχουν πρόσβαση σε σιτηρά σε παρόμοιες τιμές και σε άλλους ανταγωνιστές μας σε άλλες περιοχές του κόσμου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 65% των σιτηρών μας, των δημητριακών μας, ε, καταναλώνονται ως χορτονομές, ε, ως ε, ζωοτροφές. Συμβάλλουν δηλαδή και στην κτηνοτροφία. Οπότε η ανταγωνιστική μας θέση φαίνεται και στις εξαγωγές. Είμαστε καθαρή εξαγωγή σημαντικών ποσοστών σίτου και άλλων δευτερευόντων σιτηρών και αυτό δείχνει ότι είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί και μάλιστα όλες αυτές οι εξαγωγές γίνονται χωρίς εξαγωγικές επιστροφές, χωρίς δηλαδή δημόσιες ε, παρεμβάσεις και ε, κρατική στήριξη. Για ένα άλλο σημαντικό προϊόν, όπως το γάλα, βλέπουμε τις εξελίξεις των τιμών γάλακτος από το 2000. Η χαμηλότερη γραμμή είναι οι παγκόσμιες τιμές ε, σε ισοδύναμο γάλακτος και η πράσινη γραμμή είναι η ευρωπαϊκή τιμή γάλακτος. Η γαλάζια γραμμή είναι το δίκτυο ασφαλείας δηλαδή η τιμή για το βούτυρο και τη σκόνη και σε τι φάση παρεμβαίνουμε. Βλέπετε εδώ τις εξελίξεις του 2009. Εκεί είχαμε κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα, με πολύ χαμηλές τιμές γάλακτος. Βλέπετε όμως ότι η παγκόσμια τιμή γάλακτος το 2009 ήταν πολύ χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή τιμή. Εξαιτίας του συστήματο παρεμβάσεων που έχουμε, που ανοίξαμε και χρησιμοποίησαμε το 2009, άρχισε αμέσως μια αύξηση της τιμής γάλακτος. Διαχειριστήκαμε λοιπόν πολύ αποτελεσματικά την κρίση γάλακτος το 2009. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι οι τιμές γάλακτος στις παγκόσμιες αγορές ε, συνέκλαιναν και τώρα έχουμε την, τα 373 ευρώ τον τόνο τον Ιούλιο, τιμή Ιουλίου, που είναι σχετικά υψηλή τιμή σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε ο τομέα γάλακτος μετά την κρίση του 2009 άρχισε να σημειώνει ανωδική πορεία. Τώρα, τι είναι σημαντικό για την ανταγωνιστική μας θέση. Το σημαντικό είναι ότι εξαγάγουμε περίπου 11 με 12% της γαλακτοπαραγωγής μας. με διάφορα προϊόντα, όπως είναι το βούτυρο, το τυρί, το γάλα σε σκόνη. 11 με 12%. Και το σημαντικό είναι ότι είναι το εμπορικό ισοζύγιο και η, η η ισορροπία των τιμών γάλακτος εξαρτάται και από τις εξαγωγικές μας επιδόσεις. Έτσι συμβάλλουμε στην εσωτερική μας ισορροπία. Αλλιώς θα πρέπει, αν δεν εξάγουμε αρκετά, να μειώσουμε την εγχώρια παραγωγή γάλακτος. Έχω πολλές διαφάνειες, αλλά θα προσπαθήσω να τις περάσω γρήγορα. Για το βόηο κρέας, από το 2010 περάσαμε από τη θέση του καθαρού εισαγωγέα στη θέση του καθαρού εξαγωγέα για το χείριο κρέας και τα σχετικά προϊόντα είμαστε καθαροί εξαγωγής χείριου κρέατος και προϊόντων. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για τα πουλερικά. Τα παρόμοια κατάσταση είμαστε καθαροί εξαγωγής. Για τα αυγά το ίδιο ισχύει. Επίσης εξαγωγής τώρα για εμπορικό συζύγιο για τον ίνο. Πολύ θετικό. Το ίδιο και στο ελαιόλαδο. Είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγής παγκοσμίως σε ελαιόλαδο. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια των μεταρρυθμίσεων καταφέραμε να διασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική θέση για τους παραγωγούς μας, πολύ άνετη, και είναι σημαντικό αυτό στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Γιατί στην παγκοσμιοποίηση τα σύνορα είναι ανοιχτά. Για να κρατήσουμε λοιπόν βιώσιμη τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γεωργική παραγωγή, είναι σημαντικό να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τώρα, θα κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης. Είμαστε, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικοί στους περιοσότερους τομείς. Βέβαια, είμαστε και μεγάλη εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια ειδικά είμαστε και σημαντική εξαγωγή. Κάτι που συμβαίνει τώρα στις αγορές γεωργικών προϊόντων, εξαιτία τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση παγκόσμιες αγορέ έχουμε όλο και μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αστάθεια. Ενώ παλιά είχαμε μια κλειστή αγορά που την ελέγχαμε, τώρα με τα ανοιχτά σύνορα εισάγουμε και την αστάθεια, τη μεταβλητότητα της παγκόσμιας αγοράς. Αλλά εξαιτίας και της τεράστιας παραγωγής μας, συμβάλλουμε και σε μια σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς. Επίσης έχουμε και κάποιες διαταραχές στην αγορά. Πρόσφατα το ρωσικό εμπάργο κάποιες ασθένειες ή ε, επιζωτίες ε, ή και κακοκαιρίες, αντίξεω καιρικές συνθήκες. Αυτό που θα έχουμε, όπως είπαμε, από το χρόνο ε, θα είναι το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και επίσης και το τέλος των ποσοστώσεων στη ζάχαρη. Αλλά δεν περιμένουμε κλονισμό της αγοράς από την κατάργηση των ποσοστώσεων. Εν συντομία, ο νέος κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς ποιος είναι ο ρόλος της. Δίνει ένα αποτελεσματικό δίκτυο ασφαλείας ε, μεταξύ της δημόσιας παρέμβασης και της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Είδαμε την κατάσταση και την παγκόσμια κρίση στο Γάλα το 2009. Με το νέο κανονισμό, αυτό που κάναμε και με τη συναπόφαση, είναι να έχουμε μια πιο σταθερή κατάσταση, μια σταθερή και ασφαλή ε, κατάσταση δικαίου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κρίσεων. Έχουμε και το αποθεματικό της κρίσης, 400 εκατομμύρια με τιμές του 2011. Δεύτερη σημαντική προσπάθεια που καταβάλουμε στην ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς είναι να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς ε, να δημιουργήσουν οργανώσεις παραγωγών και να βελτιώσουν την διαπραγματευτική τους ισχύ. Γιατί ο τομέας ε, κατά ανάντι γίνεται πιο ανταγωνιστικός και πιο ισχυρός. Γι' αυτό και θέλουμε ε, να ενισχύσουμε και τους παραγωγούς στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να αποτρέψουμε την κρίση των τιμών να μεταφερθούν σε όλη, όλη την αλυσίδα των εφοδιασμών. Έχουμε και καθεστώτα ενίσχυσης για κάποιους τομείς, ε, προκυπευτικά, ίνο, ελαιόλαδο, μελισσοκομεία και ειδικά καθεστώτα για το γάλα και τα φρούτα που μοιράζονται στα σχολεία. Πρόσφατα σας στείλαμε και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μία πρόταση για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ του καθεστώτος του γάλακτος και του καθεστώτος που ισχύει για την διανομή φρούτων στα σχολεία. Άλλο σημαντικό θέμα είναι οι προδιαγραφές αγοράς στη νέα ΚΟΑ για όλα τα γεωργικά προϊόντα. Ο κανονισμός ε, δίνει ορισμούς για το τι εστί είναι στη, στη κρέας και ποια είναι τα διάφορα είδη κρέατος. Δημιουργούμε δηλαδή, αναπτύσσουμε προδιαγραφές για όλα τα στάδια της ζήτησης από τους καταναλωτές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα εξετάσουμε είναι επισήμανση προέλευσης, ε, ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε όλα τα μέτρα της αγοράς έχουμε πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, 2,7 δισεκατομμύρια. Είναι σχετικά μικρός ο προϋπολογισμός σε σχέση με τον προϋπολογισμό που έχουν οι άμεσες ενισχύσεις και από τα 2,7 δις το 1 δισεκατομμύριο θα αφιερωθεί σε προγράμματα στα απορροκυπευτικά και 1 δισεκατομμύριο στον ίνο, στις ειδικές ε, ενισχύσεις που δίνονται για τον τομέα αυτό. Τώρα, για να πάρουμε ως παράδειγμα το πρόσφατο ρωσικό εμπάργο, έχουμε τη νέα νομική βάση, το άρθρο 219, που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κατεπηγόντως μέτρα σε περίπτωση κρίσης. Και το ρωσικό εμπάργο φυσικά αντιμετωπίστηκε ως κρίση. Και άρα για τα πιο αναλώσιμα αγαθά, τα οποροκυπευτικά, αναλάβαμε άμεση δράση για να βελτιώσουμε την θέση και των οργανώσεων παραγωγών αλλά και των μεμονωμένων παραγωγών που δεν είναι μέλη ε, των ε, οργανώσεων αυτών να αποσύρουν ε, τα προϊόντα πρώιμης συγκομωδής και τις άλλες εργασίες πλην της συγκομιδής. Επίσης, δώσαμε ενισχύσεις για την απόσυρση και για την δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και προτιμήσαμε αυτό το μέτρο παρά την καταστροφή ή την αποστολή των απορροκυπευτικών στις χωματερές. Στα πλαίσια των απορροκυπευτικών είχαμε ένα μέτρο που εξαντλήθηκε σχετικά γρήγορα. Είχαμε ένα ανώτατο οικονομικό όριο που χρειάστηκε να το κλείσουμε γιατί αμέσως κατακλειστήκαμε από αιτήματα από τα κράτη-μέλη και τώρα έχουμε ένα δεύτερο μέτρο για τα απορροκυπευτικά που είναι πιο στοχευμένο και λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ε, ποσότητες που εξαγωγών προς τη Ρωσία αλλά καταρχήν καλύπτει τις ίδιες δράσεις όπως και η απόσυρση. Τώρα, ο γαλακτοκομικό τομέας, και αυτό επλήγει από το ρωσικό εμπάργο. Είχαμε ένα ειδικό καθεστώ ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα τυριά που το κλείσαμε σήμερα το πρωί γιατί και εκεί είχαμε κοινοποιήσει για τυριά που ξεπερνούσαν τα στοιχεία που είχαμε για τις εξαγωγές και αυτό και έπρεπε να κλείσουμε αυτό το ειδικό καθεστώς σήμερα το πρωί και θα δούμε αν θα το ανοίξουμε στη συνέχεια πιο στοχευμένα όμως. Στο γαλακτοκομικό τομέα όμως δεν είχαμε μόνο την ειδική αποθεματοποίηση για το τυρί, αλλά είχαμε αντίστοιχο ε, καθεστώς και για το βούτυρο και για, την, και για το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη. Και είχαμε και διεύρυνση της δημόσιας παρέμβασης ε, και της περίοδου αγοράς για το ε, βούτυρο και το αποβούτυρογμένο γάλα μέχρι τα τέλη του 2014, ενώ αρχικά ήταν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Μία άλλη πτυχή ε, όπως βλέπετε, είναι η επιτυχία που είχαν αυτές, αυτά τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά επίσης ε, πλουτίζουμε και την εμπειρία μας για τη διαχείριση των κρίσεων με τέτοια περιστατικά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα της κοινή οργάνωσης αγοράς είναι ο σχετισμός της με το δίκαιο του ανταγωνισμού κανονικά εφαρμόζεται και στην ΚΑΠ, εκτός και αν προβλέπετε κάτι, τέτοιο, εκτός και αν προβλέπετε κάτι διαφορετικό. Έχουμε κάποιες εξαιρέσεις ε, για τη ΣΚΟΑ, για παράδειγμα για συμφωνίες ε, γεωργών, για τους γεωργικού συνεταιρισμού, για πωλήσει και αποθεματοποίηση. Είναι κάτι που ισχύει εδώ και αρκετό καιρό. Και με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις θεσπίσαμε και μια καλύτερη νομική βάση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις από οργανώσεις παραγωγών σε ορισμένους τομείς είχαμε κάτι τέτοιο ήδη στο γαλακτοκομικό τομέα μετά την κρίση του 2009. Τώρα προσθέσαμε παρόμοια νομική βάση για το βόλιο, το μοσχαρίσιο κρέας, το ελαιόλαδο και τις αεροτρές καλλιέργειες. Συνεχίζουμε με ειδικά καθεστώτα σε ό,τι αφορά τον, το δίκαιο ανταγωνισμού για τα απορροκυπευτικά και τη ζάχαρη. Για τη ζάχαρη ισχύουν ειδικοί κανόνες για τη σχέση μεταξύ των παραγωγών ζαχαροτέφτυλων αφενός και της βιομηχανίας αφετέρου. Πάντως, ε, σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, καταρτίζουμε κατευθυντήρες γραμμές για τα άρθρα που διέπουν τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου και καλύτερη ερμηνεία των ε, όρων εφαρμογής αυτών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έτσι θέλουμε να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους να εφαρμόσουν καλύτερα τα άρθρα 169 έως 171. Επίσης φροντίζουμε ώστε οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να γνωρίζουν με σαφήνεια τι πρέπει να κάνουν. Ανέφερα προηγουμένως την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών. έχουμε ως πρότυπο το τομέα των προκυπευτικών. Εκεί έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα με εύρυθμη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών. Θέλουμε να το μεταφέρουμε αυτό σε όλους τους κλάδους. Επίσης έχουμε ρύθμιση της παροχής ε, τυριού και ζαμπών, ε, ένα θέμα που καλύπτεται από προστατευμένη ονομασία προέλευσης και προστατευμένη γεωγραφική έδειξη κατά έτοιμα των παραγωγών και υπό ορισμένε προποθέσει και ασφαλιστικές δικλείδε για να προστατευτούν τέτοια τυριά υψηλή ποιότητα, ή ζαμπών υψηλής ποιότητα. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν υποχρεωτικά γραπτά συμφωνητικά παράδοσης. Μερικές χώρες ήδη τα εφαρμόζουν, άλλες όχι και αφήνουν κλάδο, στον κλάδο την ρύθμιση για το θέμα αυτό. Αν τελικά τα κράτη επιλέξουν υποχρεωτικές γραπτές, ε, υποχρεωτικά γραπτά συμφωνητικά παράδοσης, έχουμε κάποια στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να υπάρχει αναρμόνιση αυτών των συμβάσεων, των συμφωνητικών παράδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε συμφωνίες και συμβάσεις ε, στον τομέα της ζάχαρης που εφαρμόζονται και κάποιες ε, εξαιρέσεις μετά το τέλος των ποσοστώσεων της ζάχαρης για το 2017. Εν κατακλείδη κάποια θέματα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε την συνήθη νομοθετική διαδικασία. Είχαμε την πρώτη εμπειρία μας από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μερικές φορές υπάρχει μια τάση να, προσ... να προσθέτουμε κάποιες λεπτομέρειες όταν μιλούμε για τον ορισμό του χυμού πορτοκαλιού ή του ορισμού του ζαμπών ή ε, τον ορισμό της μαρμελάδας. Αυτοί οι ορισμοί περιλαμβάνονται στις βασικές πράξεις και είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει. Βέβαια μπορεί να υποβάλει πρόταση, αλλά με την συνήθεια νομοθετική διαδικασία μπορούμε να φτάσουμε στην κατάσταση ώστε να θέλουμε να αλλάξουμε απλώς ένα ποσοστό, ένα τεχνικό θέμα και να χρειαστεί παρόλα αυτά να ακολουθήσουμε τη χρονοβόρα διαδικασία της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή σας, κύριε Πρόεδρε, να δείξετε εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν πρόκειται για ίσονο σημασία λεπτομέρειες και τεχνικού χαρακτήρα να τις αφήνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να την αφήνετε να αποφασίσει ελεύθερα. Αλλιώς με τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν θα γίνουμε λιγότερο αποτελεσματικοί. Τέλος, με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλες μας τις εφαρμοστικές πράξεις και να έχουμε μια σύγκληση των κατεξοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Έχουμε κυρίως, κυρίως γύρω στις 200 ε, τέτοιες νομοθετικές πράξεις για την κοινή οργάνωση αγοράς θα πρέπει να τις περιορίσουμε, να τις συμπτύξουμε σε 40. Και επ' ευκαιρία θέλουμε να τις απλουστεύσουμε κιόλα. Έχουμε εκτενείς συζητήσεις με τα κράτη-μέλη με ενδιαφερόμενους αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ομάδες που έχουμε για τις κατεξοδότηση πράξεις. Εκεί συζητούμε πώς θα απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και πώς θα ελαφρύνουμε ή θα μειώσουμε τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Επαναλαμβάνω, θέλουμε αυτές τις 200 νομοθετικές πράξεις να τις απλοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή κύριε Πρόεδρε και αν υπάρχουν ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Εννέα συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Νταντά ο πρώτος δικαιούται δύο λεπτά, οι υπόλοιποι από ένα λεπτό. Σας θερμά παρακαλώ, δικαιούται το ένα λεπτό επιπλέον ο κύριος Νταντέν γιατί είναι εισηγητής για το θέμα αυτό. Οι υπόλοιποι όμως ένα λεπτό αυστηρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό ήταν από τα πιο αμφισβητούμενα στα πλαίσια της προετοιμασίας για την κοινή αγροτική πολιτική. Ε, με αφορμή όμως το ρωσικό εμπάργο έδειξε ότι είχε τη δυνατότητα αντίδρασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα γιατί μπορέσαμε να καταστήσουμε το κείμενο αρκετά πιο ευέλικτο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση σε μια τεράστια αγορά. Εγώ ανησυχώ. Και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όταν βλέπω ποια είναι η εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής. Νέα Ζηλανδία συν 10%. Είπα 2%. Εμείς αυξάνουμε παραγωγή γεωργική, ενώ σε σχέση με την παγκόσμια αγορά έχουμε πρόβλεψη γαλακτοκομικών 15% σε ετήσια βάση. Μπροστά στην εξέλιξη αυτή της κατανάλωσης βέβαια οι τιμές δεν θα αντέξουν. Και νομίζω ότι τα μέσα που χρησιμοποιούμε, το πακέτο δηλαδή το γαλακτοκομικό, δεν επαρκούν για τη διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης γιατί στην Ευρώπη πάρα πολλοί ε, παραγωγοί όπως και στα ζαχαρότευκλα έχουν περάσει στο τέλος των ποσοστώσεων. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις σε σχέση με τα ζώα που θα περάσουν στην παραγωγή τον επόμενο χρόνο με ανησυχούν. Ποια είναι τώρα η φάση στην οποία βρίσκεται η μετάφραση των εγγράφων σε εθνικό επίπεδο. Έχετε μία αντίληψη για τις διάφορες χώρες και για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αποφασίσατε, είπατε, να μειώσετε τον αριθμό. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλεί όμως είναι η δυσκολία την οποία συναντάμε για να σεβαστείτε δηλαδή την πολιτική συμφωνία. Και αναφέρομαι στη συμφωνία για τον Ίνο που ακόμα δεν έχει καταλήξει, γενικά έχει περάσει πολλής χρόνος και ελπίζω να μην γίνει το ίδιο και με τις άλλες τέτοιες πράξεις. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ριμπέιρο. Ένα λεπτό και μόνο. Αυστηρά. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε ότι δεν περιμένετε διαταραχές από την κατάργηση των ποσοστώσεων. Μιλάμε όμως για νέα αγορά. Και μία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσε σημαντικές δυσκολίες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις ορεινές περιοχές. Στις Αζόρες παράγουμε πολύ ποιοτικό γάλα με φυσικό τρόπο. Είναι αδύνατο όμως σε μια εξόχως απόκεντρη περιοχή όπως είναι οι Αζόρες ε, να έχουμε διαφοροποίηση παραγωγής. Είναι πολύ περιορισμένη και περίπλοκη. Και φυσικά το γάλα στις Αζόρες ή το γάλα που παράγεται σε ορεινές περιοχές είναι πολύ πιο ακριβό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λέτε ότι δεν αναμένεται διαταραχή της αγοράς ή σοκ στις περιοχές αυτές από την κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Εμείς ε, στην Επιτροπή μας που είναι Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου θέλουμε μια πιο δίκαιη ε, κατανομή του βάρους στην αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Νίκολσον. Νίκολσον. Okay, chairman, I will be... Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Με μεγάλο ενδιαφέρον σας άκουσα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω πού ζείτε. Αλλά έχουν χάσει οι περιουσίες ε, οι αγρότες και τα, ο κλάδος των βοηδών τώρα τις τελευταίες 12 Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Τίποτα δεν θα μείνει αν συνεχίσουμε έτσι, ούτε στην Γαλλία, ούτε στην Ιρλανδία. Τόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Αν νομίζετε ότι τα πράγματα πάνε καλά, να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η τιμή παρέμβασης είναι ρεαλιστική αυτή τη στιγμή για τα γαλακτοκομικά? Ή μήπως θα πρέπει να έχει αυξηθεί με την τρέχουσα κατάσταση για τις ποσοστώσεις. Είπατε ότι η κατάργηση τους δεν θα έχει επιπτώσεις. Είσαστε υπεραισιόδοξος, μήπως. Ευχαριστώ κύριε Σεμπάστια. Είδαμε λοιπόν τα δύο αυτά γραφήματα σχετικά με τις τιμές των Δημητριακών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προέρχομαι από τη Βαλένσια και έχουμε επίσης πάρα πολύ υψηλή παραγωγή ε, εσπεριδοειδών. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει όμως δυστυχώς συνεχής μείωση των τιμών τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχει μια δημιουργία αίσθησης περιθωριοποίησης και ιδιαίτερα μετά από τη ρωσική κρίση. Και τα, υποτίθεται ότι θα ληφθούν μέτρα για τα οποροκυπευτικά. Για ορισμένα φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει δυνατότητα να βοηθηθούν, τα οποία δεν ξέρουμε αν τα παράγει η περιοχή. Πιστεύετε ότι το σύστημα αυτό προστασίας τους έχει ε, λειτουργήσει. Νομίζω ότι δεν το πιστεύουν αυτό οι καλλιεργητές. Ευχαριστώ. Κυρία Ριμπέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται για ανταλλαγή απόψεων με πρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Ερωτώ λοιπόν, στην παρουσίαση που έγινε για την ΚΑΠ και για τους, για τους μηχανισμούς ε, διαχείρισης και παρέμβασης στην αγορά, εκεί είναι που σημειώσαμε τη λιγότερη πρόοδο. Γιατί νομίζω ότι την ε, μάχη την κέρδισε εδώ η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και όχι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. Μας παρουσιάσατε γραφικές παραστάσεις που δείχνουν βελτίωση στο στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τότε, γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι ίδιοι γιατί πιστεύουν ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Με τις άμεσες ενισχύσεις θα δώσουμε 2% στις, στην μετάδοση της κοιτάλης ε, μεταξύ των γενναιών. Νομίζω ότι αυτό το θέμα όμω ε, είναι σχετίζεται με την αποδοτικότητα της γεωργίας. Αν υπάρχει αποδοτικότητα, πώς θα εισέλθουν οι νέοι στον τομέα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση παρά τις ωραίες γραφικές παραστάσεις που μας δείξατε. Και για το ελαιόλαδο, το 40%, το 40 του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών προέρχεται από τις άμεσες ενισχύσεις. Οπότε η αντιγωνιστικότητα που μας αναφέρατε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις άμεσες ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ παρακαλώ. Μην ξεπερνάτε το λεπτό. Η κυρία Σλάιρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε. Έχετε κάτι φυτικό να μας αναφέρετε για την ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο προσκήνιο. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Είναι οικονομικο-κοινωνική πολιτική που χρειαζόμαστε για την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρχουν οργανώσει παραγωγών, αλλά μήπως ξεχνάμε τους μικρούς φτωχούς αγρότες, γιατί δεν είναι δυνατόν να πάρουν όλες οι πολυεθνικές το κεφάλαιο και να κάνουν καταχρήσεις μεγαλύτερες από την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Είναι κρίμα που συμβαίνει αυτό. Και θα πρέπει όλοι οι κλάδοι και του βόλιου κρέας και του χειρίου κρέατος και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι να έχουν σαφήνεια για το που βρίσκονται. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόη. Grazie signor Presidente. Allora, dato che i fondi οι πιστώσεις έτσι και αλλιώς της ΚΑΠ είναι περιορισμένες για τους γεωργούς ε, και αντί να χρησιμοποιηθούν τα, τα χρήματα τα διαθέσιμα για τις κατεπίγουσες καταστάσεις και για τα εμπάργο, μήπως θα μπορούσαν ε, ε, τα προϊόντα αυτά να αγοραστούν για να ενταχθούν στην διανομή τους και στα προγράμματα τα διατροφικά στα σχολεία. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση σε ό,τι αφορά το αγροτικομικό κλάδο, όπως και ο κ. Νίκολσον, και πόσο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πιο ταχεία παρέμβαση στον γαλακτοκομικό κλάδο για να αποφύγει κρίση σε ό,τι αφορά και την κατάργηση των ποσοστώσεων. Και κατά δεύτερον, πόσο έντονε είναι οι συζητήσει μεταξύ Γενική Διεύθυνση Γεωργία και Ανταγωνιστικότητα, γιατί ξέρω ότι όταν πρόκειται για θέματα των μου είναι πολύ διαφορετικέ οι απόψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που τη θέτω από τον Αύγουστο, από τότε που έγινα ευρωβουλευτή. Τι συμβαίνει με το πρόγραμμα για το γάλα και τα απορροκυπευτικά στα σχολεία. Φαίνεται ότι η Κροατία δεν εντάσσεται, δεν επιλέξει με βάση τα ιστορικά κριτήρια. Μου υποσχέθηκε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρει κάποια λύση για να μην βρεθούν σε δυσμενή μεταχείριση τα παιδιά στην Κροατία από το πρόγραμμα αυτό για τη διανομή γάλακτος ε, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία. Επίσης, τι συμβαίνει με την προστασία του ζαμπών της Ίστριας. Είναι ένα θέμα που από το 2012. Επίσης έχουμε λουκάνικα και άλλα τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα που προσπαθούμε να επιτύχουμε για αυτά ονομασία προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Θα ήθελα λοιπόν να, γίνουν, να λεφθούν κάποια μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προστασία αυτών των τοπικών προϊόντων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και αγαπητή Επιτροπή για την παρουσίαση. Να πάρω το λόγο. Ναι, ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που βλέπουμε και νομίζω ότι ο τομέα των γαλακτοκομικών μπορεί να είναι πάρα πολύ διαγνωστικό στο παγκόσμιο προσκήνιο και όπως είπαν διάφοροι έχει υποστεί διάφορα πλήγματα σε ό,τι αφορά τα δίκτυα ασφαλείας, την εργασία. Θα πρέπει να υποστηρίξει το εισόδημα του αγρότη. Το 2015 ε, θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Ε, παρ' όλα αυτά, κάποια κρατημέλη εξακολουθούν να υποβάλλουν ε, προτάσεις για να υπάρχει κάποια διαχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει αυτό ως ενδεχόμενο ή προτιμάται μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο για να απαντήσετε, αλλά παρακαλώ εν συντομία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Σε ό,τι αφορά το γάλα. Σας έδειξα στο γράφημά μου, κύριε Νταντάν, ότι οι μέσες τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και αυτό προφανώς έχει οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτή είναι μια φυσική αντίδραση στι υψηλέ τιμέ. Σύμφωνα μαζί σα ότι οι τιμέ μπορούν να πέσουν, αλλά σε ποιο βαθμό θα επανέλθουν στα επίπεδα του 2009 είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Βλέπουμε επίσης ότι η αύξηση στην παραγωγή γάλακτος έχει απορροφηθεί από την διεθνή αγορά και από την ενιαία αγορά. Για αυτό το λόγο λοιπόν είμαι πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν το 2009, οπότε και αντιμετωπίσαμε μια χρηματοπιστωτική κρίση που επηρέασε την ζήτηση. Αν κάτι τέτοιο γινόταν ξανά ασφαλώς, θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Αλλά σε κανονικές συνθήκες πρέπει να πω ότι μάλλον θα είναι αρκετά ισορροπημένο ο τομέα του γάλακτο και η αγορά του γάλακτο. Μην ξεχνάτε ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων, γιατί Κάποιες χώρες είναι κοντά σε υπερποσοστώσεις, αλλά 20 κράτη-μέλη εξακολουθούν να παράγουν ε, κάτω από τις ποσοστώσεις και δεν έχουν τους ε, οικονομικούς όρους να αυξήσουν την, παραγωγό, την παραγωγή. Γιατί να το κάνουν λοιπόν μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015 αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διάφορες οργανώσεις παραγωγών. Στείλαμε μία έκθεση για το γάλα σε ό,τι αφορά το τι είδους οργανώσεις ε, συστάθηκαν ένα κράτος μέλος για να διαπραγματευτούν τις τιμές κτλ. Υπάρχουν λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα στον μικρό κλάδο και σε άλλους κλάδους για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Ενδεχομένω. Συμφωνείτε με τη μείωση του αριθμού σε ό,τι αφορά τις ε, εγκρίσεις στον τομέα του ίνου. Μας πήρε κάποιο καιρό το θέμα των πράξεων καταξουσιοδότησης, αλλά είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προλάβουμε να ξεκινήσει το καινούργιο καθεστώς το 2016 και όλοι οι φορείς να ξέρουν τι θα πρέπει να κάνουν στον τομέα του κρασιού σε ό,τι αφορά την κυρία Ριμπέρα και τις περιφερειακές, τις απόκεντρες περιοχές και εκεί υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί που έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να τη χάνουν διαφορετική επεξεργασία και εκτίμηση. Να έχουν διαφορετικέ δυνατότητε υποστήριξη. Αφενό. Αφετέρου, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ασφαλώ ότι δεν ε, εμποδίζουμε την ανταγωνιστικότητα όσων παραγωγών μπορούν να ανταγωνιστούν στο παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ να υπάρχει μια βιώσιμη παραγωγή. Ύστερα υπάρχει το θέμα της, ε, των τιμών παρέμβασης. Ο κύριος Νίκολσον αναφέρθηκε στο βόλιο κρέας αλλά και στα γαλατοκομικά προϊόντα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των τιμών παρέμβασης. γιατί εδώ και 30 χρόνια, ξέρετε, εργάζομαι στα αγροπτικά και έχω δει ποιες, ποια είναι τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής, της εξαγοράς. Γιατί σε κάποια στιγμή, λοιπόν, μπορεί να αγοράζουμε τέτοιες μετοχές, αλλά σε κάποια φάση θα πρέπει να βγουν αυτές οι μετοχές. Μήπως έτσι διακινδυνεύουμε παράταση της κρίσης πέρα από τα φυσιολογικά όρια. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να κρατήσουμε την ανταγωνιστική θέση που έχουμε αυτή τη στιγμή, περιορίζοντας το επίπεδο παρέμβασης και ασφαλιστικών δικλείδων. Μην ε, αντιστρέψουμε τους όρους και αρχίσουμε να τα αυξάνουμε πάλι. Και ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική αυτή για τη μείωση των τιμών ε, παρέμβασης έγινε με κάποια αποζημίωση προς τους αγρότες και αυτό αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος τους. Άρα, αφενός τους δίνουμε κάποιο ασφαλισμένο εισόδημα και από την άλλη εξασφαλίζουμε την ανταγωνιστικότητά τους. Θα ήμουν λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικό σε ό,τι αφορά την αύξηση αυτού του δίκτυου ασφαλείας γιατί θεωρώ ότι αυτό θα παρέτεινε την κρίση, θα μείωνε την ανταγωνιστικότητά μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυτροειδή, τα, τα σπριδοειδή. Θα λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά το εμπάρκο της Ρωσίας και τα σπριδοειδή. Τα σπριδοειδή λοιπόν ε, τα εξετάζουμε και αυτά σε ό,τι αφορά το ρωσικό εμπάργκο για να εξετάσουμε την, ε, τα διάφορα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας για τα σπριδοειδή σε ό,τι αφορά αυτό που είπε η κυρία Γκαρσία, σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο και το κέρδος. Ξέρουμε ότι στον κλάδο του ελαιόλαδου, του ελαιόλαδου υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που ονομάζουμε, αν θέλετε, σύγχρονες ε, δομές και παροχημένες, πιο παλιές τέτοιες υποδομές. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Τα παλιά δέντρα και ο τρόπος εσοδιάς τους οδηγεί σε χαμηλότερες ποιότητας προϊόντα και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστική μας θέση. Συμφωνώ και με τους προηγούμενους ομιλητές για να απαντήσω στην κυρία Σλέγερα ότι η μικρή οικογενειακή παραγωγή και αγρότες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας μας και θεωρώ ότι η πολιτική μας απευθύνεται, απευθύνεται και σε αυτούς. Να είμαστε όμως, να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ της ανταγωνιστικότητάς τους και μιας λύσης αποδεκτής για μας. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να σταματήσω, να σταματήσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Αν κάποιος δεν έλαβε απάντηση, μπορεί να στείλει γραπτό στην ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περνάμε στο επόμενο θέμα, τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, ανάπτυξη υπαίθρου. Το λόγο έχει ο, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Μιχάηλ Ντουμίτρου. Και στον επόμενο γύρο ερωτήσεων θα είναι μονόλεπτες οι ερωτήσεις. Άλλωστε νομίζω ότι είναι λιγότερο επίμαχο και αφιλεγόμενο το θέμα, οπότε θα έχουμε και λιγότερους ομιλητές φαντάζομαι και συντομότερη συζήτηση. Αυτή ήταν άλλωστε η λογική, ότι να ακούσουμε πρώτα τα πιο φλέγοντα θέματα των άμεσων ενισχύσεων και της κοινή οργάνωσης αγοράς και σε αυτά να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Τώρα για την αγροτική ανάπτυξη και τον οριζόντο κανονισμό έχουμε λιγότερο χρόνο. Παρακαλώ κύριε Ντουμίτρου. μίλησε για να σας δώσω το χρόνο να εγκατασταθείτε. Παρακαλώ σας ακούμε κύριε Διευθυντά. Δέκα λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας. Κυρίε και κύριοι, θα προσπαθήσω σε 10 λεπτά να σας δώσω κάποια βασικά στοιχεία τη πολιτική για τη ανάπτυξη του Υπέθρου για την περίοδο 2014-2020. So, first of all, I just... Καταρχάς, για να σας παρουσιάσω εν συντομία τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχει η πολιτική αυτή στη νέα περίοδο. Ο βασικός στόχος του αγροτικού κλάδου είναι η παραγωγή τροφίμων. Ωστόσο, η γεωργία συμβάλλει όλο και πιο πολύ στην παραγωγή ενέργειας και βιομάζας ιδιαίτερως. Αν θέλουμε όμως να διατηρήσουμε το δυναμικό της γεωργίας και στο μέλλον, θα πρέπει να φροντίσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων και να υπάρξει βιώσιμη διαχείριση των εθνικών πόρων, ιδιαίτερως ε, του εδάφους και του ύδατος, του νερού. Οι αγρότε όμως όλο και πιο πολύ αντιμετωπίζουν τι συνέπειε της αλλαγής του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τους παρέχουμε και μέτρα και δράσεις απάλυνσης ε, του φαινομένου αυτού. Η ευρωπαϊκή κοινωνία δίνει μεγάλη σημασία στη διατηρήση των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας. Αυτό όμως δεν έχει μηδενικό κόστο. Θα πρέπει λοιπόν να αποζημιώσουμε του αγρότε που παρέχουν αυτά τα δημόσια αγαθά κοινότητες της Υπέθρου έχουν μεγάλη ιστορία και δίνουν μεγάλη σημασία στον πολιτισμό και στις αξίες τους. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να γίνονται χωρίς να διατηρείται η οικονομική βιωσιμότητα του αγροτικού κλάδου. Και ε, ε, στο σύνολο, θα πρέπει, στο σύνολο της θα πρέπει να κοιτάξουμε και στο οικονομικό-κοινωνικό ε, πλαίσιο το θέμα της γεωρικής ανάπτυξης η πολιτική ανάπτυξη της Πέτρου πώς αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε όλους τους στόχους που προβλέπονται στο νέο κανονισμό για την ανάπτυξη της Πέτρου αλλά θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στις έξι προτεραιότητες για την ανάπτυξη της υπαίθρου για τη νέα προγραμματική περίοδο. Οι προτεραιότητες αυτές είναι κάτι που διαμορφώνεται και σε τομείς εστίασης, οι οποίοι στη συνέχεια περιλαμβάνουν κάποια μέτρα. Καταρχάς, λοιπόν, προτεραιότητα μεταφορά γνώσης και καινοτομία. Και θέλουμε, λοιπόν, οι αγρότες να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία, στις ε, νέους ιδέες, σε νέους τρόπους. Αυτό γίνεται μέσω ανταλλαγή, ε, μέσω εκπαίδευση, μέσω συμβουλευτική. Ε, προς τους γεωργούς μέσω ε, πιλωτικών προγραμμάτων δικτύωσης των ε, αγροτών. Δεύτερη προτεραιότητα της ανάπτυξης της Πέτρου είναι η βιωσιμότητα όλων των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλες τις περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υποστηρίξουμε την αηφορία. Για παράδειγμα, η προώθηση της επικοινωνία των νέων επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος προκειμένου να διατηρείται ο ενθουσιασμός των γεωργών και να υπάρξει για ανανέωση των γενεών. Πολύ σημαντικό αυτό για να διατηρηθούν οι περιοχές της υπαίθρου μας. Τρίτη προτεραιότητα, καλύτερη ενσωμάτωση της αλυσίδας των τροφίμων, αλλά και παροχή μέσων για την ε, διαχείριση των κινδύνων και για την ευημερία των ζώων. Θέλουμε οι αγρότες να ενταχθούν καλύτερα στην αλυσίδα των τροφίμων και θέλουμε να αυξάνουν τα κέρδη τους. Αυτό πώς μπορούμε να το πετύχουμε, ε, Μικράντα την αλυσίδα εφοδιασμού, παραγωγής τροφίμων, υποστηρίζοντας ε, τις τοπικές αγορές και θέλουμε επίσης να προστατεύσουμε τους γεωργικούς, να τους δώσουμε πιο πολλά μέσα και εργαλεία για να προστατεύονται κατά των κινδύνων, κατά των κυρικών συνθήκων, κατά των ασθενειών των, ε, του αίματος, των επιζώτιων, καλύτερες ασφάλειες. Η μέσω ανάπτυξης κοινων ταμείων, μέσω ανάπτυξης μέσων για σταθεροποίηση του εισοδήματός τους. Τέταρτη προτεραιότητα, τα οικοσυστήματα εδώ θέλουμε να καλυφθεί η βιοπικιλότητα, η προστασία του νερού και του εδάφους. Όσοι γνωρίζετε τα μέτρα για το αγροπεριβάλλον, ξέρετε ότι οι αγρότες που μπαίνουν σε καθεστώς ε, εθελοντικών δεσμεύσεων πάνω από το προβλεπόμενο επίπεδο αποζημιώνονται για τα δημόσια αγαθά που παρέχουν. Εδώ λοιπόν στην προτεραιότητα αυτή παρέχουμε ενισχύσεις για να διατηρούνται οι γεωργικές δραστηριότητες σε περιφέρειες που έχουν φυσικούς περιορισμούς. Πέμπτη προτεραιότητα. Αποδοτικότητα των πόρων και ε, μετάβαση σε μια ανθεκτική οικονομία στον τομέα της γεωργία και τη δασοκομεία. Εδώ καλύπτονται πέντε διαφορετικοί τομείς ε, ενέργειας, αποτελεσματική χρήση νερού και εδάφου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειονέργεια, μείωση των αερίων ε, του θερμοκηπίου και τη αμμονία και διατήρηση του άνθρακα. Τέλος. Η έκτη προτεραιότητα έχει να κάνει με την κοινωνική συμπερίληψη και τη μείωση της φτώχειας ευημερία του κόσμου που ζει στην Ήπεθρο. Είναι σημαντικό που αυτή η προτεραιότητα μπορεί να παρέχει, να περιλαμβάνει και τις τηλεπικοινωνίες, την παροχή υποδομών, ε, ευρωζωνικές συνδέσεις, ε, δημιουργία θέσεων εργασία, να βελτιώσει την ε, ισότητα στην Ήπεθρο. Και στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε και την προσέγγιση LEADER που έχει πλέον 20 ετή ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα, κάθε κράτος μέλος θα κληθεί να αποφασίσει και να επιλέξει τέσσερις τουλάχιστον από τις έξι αυτές προτεραιότητες για να μπορέσει να καταλήξει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Πόσα χρήματα λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας για να τα πετύχουμε αυτά. Πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησε για 95,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Αυτό σε τρέχουσες τιμές. Και το 2, σε τιμές 2011 αποτελεί ε, ποσό 85 δισεκατομμυρίων. Δεν είναι μόνο αυτά τα χρήματα που έχουμε στην διάθεσή μας ασφαλώς. Έχουμε και εθνικές χρηματοδοτήσεις και περιφερειακές χρηματοδοτήσεις από περιφερειακές αυτοδιοίκησεις και επίσης και σε μερικές περιπτώσεις και συνεισφορά από τους ιδιώτες. Είναι συγχρηματοδοτούμενη η πολιτική, η πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Το τονίζω αυτό και ξέρετε ότι, για παράδειγμα, ε, οι φάκελοι αυτοί, τα προπολογισμοί που προβλέπονται για κάθε χώρα. Στις χώρες όπου υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα εκτελούνται από τις εθνικές αρχές. Και θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι τα ποσά αυτά υποβάλλονται σε, υποβάλλονται σε συγκεκριμένους όρους και αυτό δεν σημαίνει ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις, ε, ε, τις προτάσεις τις επόμενα τρία χρόνια μετά από το χρόνο που αναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις. Ιδάλλως χάνουν τα χρήματα αυτά για το εθνικό πρόγραμμα και πάνε ε, επιστρέφουν στον ευρωπαϊκό προλογισμό. Ε, εδώ, στην τρέχουσα περίοδο, ισχύει ο κανόνας νήσιν 2, όχι νήσιν 3. Τα κράτη-μέλη, λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, έχουν ε, την δυνατότητα να προτείνουν εθνικά προγράμματα, περιφερειακά προγράμματα ή συνδυασμό εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Και κάποια κράτη-μέλη αν έχουν ε, ε, περιφερειακά προγράμματα, προτείνουν εθνικά προγράμματα για κάποια άλλα ζητήματα. Και επίσης μπορεί να προτείνουν τα κράτη-μέλη και ένα εθνικό πλαίσιο για το πώς θα σχεδιάζονται τα περιφερειακά προγράμματα. Άρα σήμερα έχουμε 118 προγράμματα Ανάπτυξη της υπαίθρου που πρόκειται για αύξηση σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο και κάποια αποφάσισαν να εφαρμόσουν πιο πολλά προγράμματα ή να περάσουν σε περιφερειακό επίπεδο και αναφέρουμε στη Γαλλία, στην προκειμένη περίπτωση. Πώς θα τα πετύχουμε λοιπόν όλα αυτά. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω όλο το εύρος των μέτρων που, παρου... που περιλαμβάνοντα τον κανονισμό για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διεξαγάγουν μια ανάλυση για να βρουν τα δυνατά σημεία του και τι αδυναμίε του. Και μετά θα πληθούν να επιλέξουν προτεραιότητες, να επιλέξουν στόχου, να επιλέξουν ένα μείγμα μέσων και να προβλέψουν και χρηματοδότηση. τρεις κατηγορίες. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ε, πληρωμές για τη διαχείριση της γης και συνεργασία. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική σε τοπικό επίπεδο μέσω του Leader ή μέσω άλλων προγραμμάτων συνεργασίας. Όπως ανέφερε και ο Γενικός Διευθυντής μου, είμαστε σε στενή συνεργασία με τα άλλα επενδυτικά και γεωργικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να καταρτήσουμε μια συμφωνία εταιρική σχέση, την οποία θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσει στη διαδικασία κατάρτιση προγραμμάτων. Αυτό όμω δεν αποτελεί και το τέλο τη ιστορία αυτή. Ε, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα προγράμματα για να δούμε κατά πόσο επιτυχάνονται οι στόχοι. Και αυτό θα το κάνουμε το 2017-2019. Τελευταίο σημείο, συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε σε αυτή τη διαδικασία σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε από Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, ε, Επιτροπή στην προγραμματική ε, φάση συνεργαζόμαστε με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με του αγρότες, με τις εθνικές τοπικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δεν αποτελεί και το τέλος της ιστορίας, ακόμα και για τη φάση του ελέγχου και τη επιτήρησης υπάρχει συνεργασία μεταξύ διάφορων φορέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και να απαντήσω ευχαρίστω στις ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Διαπιστώσατε ότι είναι σχετικά ελαφρές, ελαφριές ε, οι παρουσιάσεις. Είναι πιο εικονικές, είναι εικαστικές θα έλεγα. Έχουν ε, πολλές, πολλούς πίνακες και φωτογραφίες. Ο κύριος Νταντά, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μία απλούστατη ερώτηση έχω να κάνω. Γιατί πλησιάζουμε στα τέλη του 2014. Πόσα περιφερειακά προγράμματα έχετε λάβει από τα 118. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση Έμαθα ότι στείλατε απαντήσεις σε εθνικές και αρχές και έχω την αίσθηση ότι αυτά που στερηθήκατε από τον κανονισμό τα παίρνετε πίσω από την εκτέλεση. Και μιλήσατε για τη λήψη υπόψη του περιβάλλοντος. Αυτό όμως ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της πολιτικής συμφωνίας και σας κρύω το κόδωρο του κινδύνου. Αν οι ευρωβουλευτές διαπιστώσουν πρόβλημα στη διαμόρφωση των κειμένων, την επόμενη φορά θα είμαστε πολύ πιο σχολαστικοί και θα στριμώξουμε πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιορίζοντας το περιθώριο λιγμών τη. Είχαμε μεταξύ μα ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Θα ήθελα να το τηρήσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Γιάρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία διαπίστωση, δύο ερωτήσει. Διαπίστωση. Πιστεύω ότι είναι καλό το γεγονός ότι διαμορφώνεται η Ήπετρος με ε, αγροτικό τρόπο για την αγροτική πολιτική και όχι σε άλλες, προς άλλες κατευθύνσεις. Κατά δεύτερον, είπατε ότι όλα τα ταμεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία, κατά μία ομπρέλα. Καλό είναι αυτό, αλλά ποιος θα φροντίσει να υπάρχει σε λιγότερη γραφειοκρατία. για να μην χαθούν τα καλά στοιχεία της μεταρρύθμισης και να μην χανόμαστε στη γραφειοκρατία είναι κάποιος που ε, φροντίζει να συνενωθούν όλα αυτά, αλλά και να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος, να μην αυξηθεί κιόλα. Τελευταία ερώτηση. Μας ε, είπατε ότι το, μάλλον ε, αποδείχθηκε ότι το πρασίνισμα ε, θα έπρεπε να είναι στη δεύτερη πυλώνα. Για μένα είναι αυτό αυταπόδεκτο. Εσείς συμφωνείτε, μπορείτε να το να μας πείτε την άποψή σας. Σας ευχαριστώ, η κυρία Πετήρ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Η Κροατία υπέβαλε το πρόγραμμά τη για την αγροτική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε κάποια περαιτέρω επεξεργασία και νομίζω ότι το καλοκαίρι υπευλήθηκε το συμπληρωματικό σχέδιο. Αλλά για φέτος φαίνεται ότι χάσαμε στην Κροατία τα κονδύλια από την αγροτική ανάπτυξη. Αυτή τη φορά θα αξιολογήσετε θετικά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Κροατίας και πότε θα μπορέσει η Κροατία να αξιοποιήσει τα κονδύλια που δικαιούται. Ευχαριστώ. Κυρία Γκουιλέρα, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση για την ανάπτυξη πέθρου. Βέβαια, πρωταρχικός μας στόχος είναι η υποστήριξη των νέων. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο να προσελκύσουμε τους νέους στη γεωργία. Στο προηγούμενο όμως πλαίσιο που είχαμε δεν λειτουργήσαν οι ενισχύσεις και δεν προσήλκησαν νέους στην γεωργία. Εγώ από την Ανταλουσία έχουμε σημαντική γεωργία και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο μεταποίησης. Δεν μπορέσαμε όμως να εφαρμόσουμε τις ενισχύσεις του προηγούμενου πλαισίου για να περιλάβουμε πολύ περισσότερους νέους στη γεωργία και για την άρδευση. Γιατί ε, δεν ε, δίνεται μέτρα και για την ε, μετατροπή παρά μόνο για τον εξυγχρονισμό της άρδευσης. Ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ θα ήθελα να μάθω πόσα σχέδια έχετε εγκρίνει από τα κράτη-μέλη και πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Γιατί είναι αρκετά επαχθές το έργο Θέλουμε να εφαρμοστούν τα σχέδια σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Πέντε ερωτήσεις σας υποβλήθηκαν, μισό λεπτό για την κάθε απάντηση. Έχετε δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πρώτον, η διαδικασία είναι συνεχιζόμενη. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, παίρνουμε τις προτάσεις τους, τις αναλύουμε, στέλνουμε επιστολές παρατήρησης και αφού πάρουμε απαντήσεις περνάμε στη διαδικασία αποδοχής. Μέχρι τώρα πήραμε 112 ή 118 μάλλον προτάσεις. Έχουμε πάρει τις 112 και περιμένουμε εν πάση περιπτώσει τις υπόλοιπες 6 τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα για την έγκριση του προγράμματος δεν έχουμε εγκρίνει κανένα. Γιατί τα πήραμε λίγο πριν το καλοκαίρι. Και γιατί πρέπει να υπάρξει καταρχάς η συμφωνία της εταιρική σχέσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 16 μέχρι τώρα από τις 28 συμφωνίες εταιρική φύσεως. Λοιπόν, πρέπει να αναλύσουμε τα σημαντικά αυτά έγγραφα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έχουμε μια προθεσμία για να στείλουμε τις παρατηρήσεις μας ε, τριών μηνών και θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις. Αν οι απαντήσεις είναι καλές και δίδουν πραγματικά τα στοιχεία που θέλουμε, περνάμε γρήγορα στην υιοθέτηση του προγράμματος. Τώρα για την εφαρμογή. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε αυτά τα οποία λέει ο κανονισμός. Προφανώς προσπαθούμε εμείς να βάλουμε στο πρόγραμμα ένα φιλόδοξο επίπεδο στόχευσης. Αλλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις. Τέλος, για την απλούστευση και το διοικητικό άχθος. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία απλουστευτικά στα πλαίσια της νέας πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Καταρχάς ευθυγραμμίζουμε κάποια στοιχεία με τους κανονισμούς των άλλων ταμείων, Απλωστεύουμε τις διαδικασίες σε επίπεδο πολιτικών, αλλά το θέμα είναι τι θέλουν τα κράτη-μέλη να προτείνουν στα προγράμματα αυτά και αν θέλουν να κρατήσουν τα προγράμματα αυτά σε μια κατάσταση όχι ιδιαίτερα περίπλοκη. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Πρώτον το τι είναι γραμμένο στο πρόγραμμα και έγινε δεκτό από την Επιτροπή και τι κάνουν τα κράτη-μέλη από την άλλη. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με τα κράτη-μέλη και το κάνουμε αυτό για να απλουστεύσουμε και από τις δύο πλευρές, γιατί αλλιώς ο τελικός θα θέλετε αυτός που θα ωφεληθεί από τη διαδικασία θα καθυστερήσει. Συνεργαζόμαστε και με την Κροατία. Στην αρχή όπως και με άλλα κράτη-μέλη είχαμε ξεκινήσει κάποιες ανεπίσημες μορφές διαδικασίας Τώρα έχουμε περάσει στις επίσημες συζητήσεις. Για τους νέους γεωργούς, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, μπορώ να απαντήσω. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία τα οποία μπορούν να καταστήσουν τους νέους γεωργούς να ενδιαφερθούν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής. Έχουμε καλύτερες δυνατότητες εμπλοκής με τον πρώτο πυλώνα και μπορούμε να στηρίξουμε επίσης και μέσω συμβουλών, μέσω κατάρτισης έτσι ώστε να, ζητήσουμε, να πείσουμε τους γεωργούς αυτούς να κάνουν αιτήσει για την εφαρμογή των μέσων. Ευχαριστώ και περνάμε στην τελευταία παρουσίαση από τον κύριο Μέγκελε που είναι αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ε, της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη για τον οριζόντιο κανονισμό και εσείς ένα δεκάλεπτο έχετε και μετά ερωτήσεις ενός λεπτού. Παρακαλώ κύριε Μέγκελε, έχετε το λόγο.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 Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέραν των τεχνικών λοιπόν, αφού τα λέξαμε, μπορώ να ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας τον οριζόντιο κανονισμό, το τέταρτο έγγραφο δηλαδή που υιοθετήθηκε στη φετινή περίοδο, που ξεκίνησε το 2013 μάλλον, προετοίμασα λίγες διαφάνειες για σας, υπάρχουν περισσότερες διαφάνειες που είναι και αυτές στη διάθεσή σας και οι οποίες είναι λεπτομερέστερες και σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Τι θα βρείτε τι και πού στο έγγραφο. Ίσως κάποια από αυτά να σας φανούν περίπλοκα και τεχνικά και γι' αυτό δεν τα παρουσιάσω στην αρχή. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του οριζόντιου κανονισμού είναι η μετατροπή των πολιτικών προτεραιοτήτων σε πραγματικότητα, δηλαδή η διαχείριση και εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής. Επίσης, αντικατοπτρίζει και τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν αποφασιστεί εκτός Γεωργίας. Τρία βασικά έγγραφα, τα οποία προέρχονται από τις ε, διαδικασίες λήψης απόφασης στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος. Καταρχάς, ο κανονισμός των κοινών προβλέψεων που περιλαμβάνει πολλούς, πολύ συγκεκριμένους κανόνες για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπάρχει ο γενικότερος δημοσιονομικός κανονισμός, ο οποίος έχει αλλάξει αρκετά και έχει επηρεάσει φυσικά τον οριζόντιο κανονισμό και υπάρχει και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο το ίδιο το πλαίσιο χαρακτηρίζει θα έλεγα τον κανονισμό αυτό και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Στόχοι τώρα του οριζόντιου κανονισμού είναι βασικά τριών ειδών. Πρώτον θέλουμε να πετέχουμε μια καλύτερη εφαρμογή και μια καλύτερη διαχείριση της ΚΑΠ βελτιώνοντας και ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες. Θέλουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις ευρωπαϊκές πιστώσεις. Αυτός είναι ένας στόχος παλαιός σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Και τέλος θέλουμε να ε, σταθεροποιήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να περιλαμβάνονται δηλαδή αρκετά έγγραφα τα οποία ήταν κατανεμημένα σε διαφορετικά σημεία των νόμων των κοινοτικών. Ε, ποιες είναι τώρα, ποια είναι τα μέσα αυτά, τα εγκάρσια θα έλεγα, στα πλαίσια του οριζόντιου κανονισμού. Καταρχάς οι κανόνες ε, διαχείρισης για την Επιτροπή σημαντικό αλλά και για τα κράτη-μέλη στις καθημερινές τους ενασχολήσεις με τους γεωργούς σχετικά με τη χρηματοδότηση των μέτρων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Διαχείριση και ελεγκτικά συστήματα στα κράτη-μέλη εκαθάριση λογαριασμών στο σύστημα του clawback, δηλαδή ανάκτηση χρημάτων που έχουν δαπανηθεί αδικαιολογήτως, ανακτήσεις ποσών, κυρώσεις, πρόστιμα, παρακολούθηση, διαφάνεια και άλλα θέματα τα οποία δεν παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι το Άιαξ έχει παρουσιαστεί από τον κύριο Μπάσκου και δεν θα πω πολλά πράγματα για αυτά και το ίδιο ισχύει επίσης και για τις διάφορες μορφές συμμόρφωσης. Τώρα, ποιος κάνει τι στα πλαίσια αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Υπάρχουν δύο βασικοί εταίροι στα πλαίσια της εφαρμογής και διαχείρισης της ΚΑΠΑ. Από τη μία τα κράτη-μέλη, με τις ε, υπηρεσίες πληρωμών, τους οργανισμούς πληρωμών και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε τα δύο για να καταλάβουμε το ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Εξ αριστερών έχετε τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες πληρωμών, τους οργανισμούς πληρωμών. Ασχολούνται άμεσα με τους γεωργούς που ζητούν επιδότηση, ενίσχυση, ελέγχουν τα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί πληρωμών δίδουν τα χρήματα. Εκ δεξιών βλέπετε ότι τα κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες αυτές δηλώνουν τις δαπάνες τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει το αν οι ισχυρισμοί είναι ορθοί και γίνονται εκ των υστέρων πολλές φορές και έλεγχοι, οπότε εκεί ίσως πιθανώς να υπάρχουν και δημοσιονομικές διορθώσεις όταν έχουν παραβιαστεί οι κοινοτικοί κανόνες είναι το θέμα της εκαθάρισης ε, και πιστοποίησης των λογαριασμών. Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Ε, υπόθηκε εδώ ότι από τη μία έχει σημασία να υπάρξει ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο σφαίρες σχετικά με την ε, κατανομή των ευθύνων ταυτόχρονα. Έχει υποθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται και να στηρίζει τα κράτη-μέλη και να καθορίζει τον τρόπο που εφαρμόζουν τις πολιτικές. Τα τα δύο δείχνουν τη δυσκολία και την περιπλοκότητα της διαδικασίας. Βρισκόμαστε στα πλαίσια της μικτής διαχείρισης. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κάνουν μεν δύο διαφορετικά πράγματα. Από την άλλη υπάρχει αλληλοεπίδραση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει σωστή οργάνωση μεταξύ τους. Τώρα για η πιο αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση της κοινή αγροτικής πολιτικής γενικά θα έλεγα δεν έχει αλλάξει η δημοσιονομική διαχείριση στον οριζόντιο κανονισμό. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Πρώτον, είναι το λεγόμενο μέσο δημοσιονομικής λιτότητας, πειθαρχία. Αυτό διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα όρια. Τα όρια αυτά καθορίζονται από το, από το πολιετές δημοσιονομικό και πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όταν προβλέπεται οι δημοσιονομικές ανάγκες να είναι υψηλότερες από τις πιστώσεις που είναι διαθέσιμες, τότε γίνονται κάποιες προτάσεις προς τις νομοθετικές υπηρεσίες στο νομοθετικό επίπεδο και αυτή θα κρίνει αν θα υπάρξουν αλλαγές. Αυτό το μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιηθείτε ε, σε αιτήσια βάση για να ε, βρίσκονται και χρήματα για το λεγόμενο ταμείο ε, κρίσης ή αποθεματικό κρίσης. Προβλέπεται να φτάσουν τα 400 εκατομμύρια σε τιμές του 11. Αυτό σημαίνει για το 2015 ότι θα έχουμε 433 εκατομμύρια τα οποία θα είναι διαθέσιμα για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων. Το αποθεματικό αυτό λειτουργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κινητοποιείται η δημοσιονομική πειθαρχία όταν υπάρχουν μειώσεις από τις άμεσες ενισχύσεις τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό. Αν δεν χρειάζονται μέτρα για αντιμετώπιση κρίσεων, τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται, θα έλεγα, στους γεωργούς τον επόμενο χρόνο. Ποιο είναι το πλεονέκτημα τώρα αυτού του διπλού συστήματος. Κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος και να περιμένει ότι σε ένα δεδομένο χρόνο μια κρίση η οποία να εντάσσεται σε αυτά τα κριτήρια θα υπάρξει. Τα χρήματα θα χάνονται στο τέλος του χρόνου, ε, χάνονταν μάλλον στο τέλος του χρόνου. Τα χρήματα όμως αυτά τώρα θα επιστρέφονται στους γεωργούς τον επόμενο χρόνο. Αν, αν, αν υπάρχει ανάγκη για τη χρήση όμως των ποσών του αποθεματικού, τότε θα χρησιμοποιούνται και θα καταναλώνονται και η επιστροφή των χρημάτων αυτών μέσω των άμεσων ε, πληρωμών ενισχύσεων δεν θα ισχύει. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς θα χρησιμοποιείται το αποθεματικό της κρίσης, περιλαμβάνεται στον αρμόδιο κανονισμό. Να αναφερθώ τώρα στο θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Εδώ υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις δημοσιονομικές οι οποίες προβλέπονται και στον οριζόντιο κανονισμό. Δεν υπάρχει βέβαια δυνατότητα διπλής χρηματοδότησης γύρω από το screening της ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχει αυξηθεί σε 3% αυτό έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου ενδιάμεσες πληρωμές μπορεί να καλύψουν το 95% του προγράμματος changed into N which... και από το M 2 περάσαμε στο M 2, δηλαδή ανάμεσα στις, ε, στην εγγραφή συγκεκριμένων πιστώσεων και στη χρήση ε, των ποσών αυτών από το κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να μεσολαβούν περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ στον προηγούμενο κανονισμό τα χρόνια αυτά ήταν δύο. Τώρα, για να υπάρξει αποδέσμευση των πιστώσεων αυτών. Αναφέρθηκα λοιπόν στα, διαχειριστικά συστήματα, στο Ajax. Το σύστημα αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρξει σωστή διαχείριση του συνόλου των 7,8 εκατομμυρίων πρόσφατα ετοιμάτων για άμεσες ενισχύσεις. Αυτό το καλύπτουν φυσικά οι, οργανισμοί πληρωμών. Υπάρχει έλεγχος μεταξύ των οποίων των μορφών ελέγχου υπάρχουν και οι αεροφωτογραφίες που επαληθεύουν τις επιλέξιμες και μη επιλέξιμες περιοχές. Το σύστημα αυτό δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Από το 2018 θα υπάρξει ένα ενδιάμεσο επίπεδο για το greening, ιδιαίτερα για τις περιοχές υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει το συμβουλευτικό σύστημα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπήρχε στο παρελθόν, τώρα έχει διευρυνθεί η εμβέλειά του. Έχουν υπάρξει νέα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν, ιδιαίτερα τα θέματα διαχείρισης ε, και σε σχέση ε, με το τι λένε συγκεκριμένοι κανονισμοί για την ε, έλογη χρήση των farm Των φυτοφαρμάκων και τη χρήση των υδάτινων πόρων και διάφορες άλλες επιμέρους ε, ρυθμίσεις. Τώρα έλεγχη και πρόστιμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν ελέγχου φυσικά πριν πληρώνουν ε, τα χρήματα αυτά, είτε άμεσα είτε με διαφορετικό τρόπο. Οι βασικοί κανόνες για τους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται στον οριζόντιο κανονισμό Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, πράξεις και επίσης και κατεξουσιοδότηση πράξης. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόστιμα. Να αναφερθώ σε ένα πρόστιμο το οποίο είχε παρουσιάσει αρκετά θέματα προσυζήτηση στην μεταρρύθμιση αφορούσε το πρασίνισμα, το greening. Πρόκειται για μια μεταβατική φάση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Τα δύο πρώτα χρόνια στο συγκεκριμένο θέμα του greening δεν θα υπάρξουν πρόστιμα και θα υπάρξει δυνατότητά τους από τον τρίτο χρόνο και μετά που μπορεί να φτάνει το 25%. Ένα άλλο μέσο ε, ακύρωσης της διαδικασίας πληρωμή. Αν δούμε ότι ένα πρόγραμμα δεν εξελίσσεται σωστά σε ένα κράτος μέλος, ζητάμε από το κράτος μέλος ένα πρόγραμμα δράσης. Αν η αδυναμία αυτή δεν αντιμετωπιστεί ορθά, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει ένα τμήμα των πληρωμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις μειώσει. Ή να πει ότι θα υπάρξει μια εκτονιστέρων απόφαση στα πλαίσια της εκαθάρισης ε, των λογαριασμών. Ε, κάποια μέσα εκτονιστέρων, δηλαδή συμπληρώνονται. Τέλος υπάρχει μια ρήτρα για την εφαρμογή σε επίπεδο αποκέντρωσης αυτό αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε ορισμένες χώρες οι οποίες είναι αρκετά περιφερειοποιημένες όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο που ενδιαφέρονται σε για αυτήν την περιφερειοποίηση. Τώρα, καλύτερη προστασία των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ανακτήσεις ποσών. Έχουμε κάνει κάποια βήματα ευθυγραμμίζοντας τις διαδικασίες θα σας παραπέμψω σε λεπτομέρειες στις επιπλέον διαφάνειες. Έχουν υπάρξει νέα συστήματα παροχής διασφαλίσεων, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν επιπλέον μέσα ελέγχου της ορθότητας των μέσων διαχείρισης και αυτό θα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Να έχουμε επαρκείς διαβεβαιώσεις δηλαδή. Και τέλος η διαδικασία όπως είπα εκαθάρισης των λογαριασμών το οποίο βρίσκεται εκεί έτσι ώστε αν υπάρξουν ε, δαπάνες μη τεκμηριωμένες τα χρήματα να ανακτώνται. Η διαδικασία αυτή έπαιρνε πάρα πολύ καιρό, τώρα τη συντομεύουμε γενικά Τώρα θα πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση μέσα σε δύο χρόνια. Και τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται για καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις ε, ορίζονται πλέον και στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, όχι μόνο στον κανονισμό. Υπάρχει επίσης ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης και παρακολούθησης το οποίο δείχνει ότι η πολιτική σε ένα χρονικό διάστημα έχει αποδώσει και αν όχι γιατί δεν έχει καλά αποδώσει τα αναμενόμενα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Στον 834 έχει καθοριστεί ένα, μια σειρά δίκτων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μέσων της κοινή αγροτικής πολιτικής στο τέλος, πριν το τέλος μάλλον του 18 θα παρουσιάσει μια έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνει το ίδιο ανά τέσσερα έτη. Τέλος, ένα άλλο θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι η διαφάνεια σχετικά με τα ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί δηλαδή προς αυτούς οι οποίοι δικαιούνται, τους δικαιούχους. Ενθυμίστε ότι το σύστημα αυτό είχε ακυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άλλαξε, μεταρρυθμίστηκε για να καλυφθούν οι αδυναμίες που είχε εντοπίσει το, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα θα δημοσιοποιείται το όνομα του δικαιούχου, ο Δήμος ή η κοινότητα, τα ποσά που παίρνει και τι χώρες φυσικά. Έτσι λοιπόν θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των πιστώσεων και θα έχουμε καλύτερες εικόνες για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Η πρώτη δημοσίευση με βάση τους νέους κανόνες που θα καλύπτει το 14 θα δημοσιευθεί το 15. Λοιπόν, είναι μια σύντομη παρουσίαση ενός κανονισμού λεπτομερέστατου και περίπλοκου θα έλεγα, αλλά νομίζω ότι είναι βασικό για τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν ε, τον κανονισμό αυτό με σωστό τρόπο. Είμαι έτοιμος για να δεχθώ ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ε, έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο μας. Ευτυχώς έχουμε μόνο μία ομιλήτρια στο γύρο αυτό, η κυρία Μαγκίνες που θα ξεκινήσει και θα ολοκληρώσει. Α, όχι, βλέπω και την κυρία Μόη που ζήτησε το λόγο. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, πολύ χρήσιμη, για να θυμηθούμε κάποιες λεπτομέρειες που είχαμε συμφωνήσει, ιδιαίτερα για το πρασίνισμα, το greening. Είπατε ότι το 2018 και 2020 θα προσθεθεί ένα νέο στρώμα στο σύστημα για να γίνει καλύτερη διαχείριση του πρασινίσματος. Τι σημαίνει αυτό, ότι το παρόν σύστημα δεν ελέγχει επαρκώς το, το και αν ο έλεγχος γίνεται με επιθεωρήσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τα πρώτα δύο χρόνια και δεδομένου ότι τα πρόστιμα θα εφαρμοστούν μόνο το 2017. Τι σημαίνει ότι δεν έχουμε με το ισχύον σύστημα αρκετό έλεγχο του greening, του πρασινίσματος. κυρία Μόη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ότι στην Ιταλία αυτά τα, αυτές οι ευρωπαϊκές πιστώσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου πολύ συχνά χρησιμοποιούνται με παράνομο τρόπο και πάρα πολλές φορές οι ελεγκτές συμμετείχαν στην απάτη και αυτό δημιούργησε ένα πολιτικό πελατειακό σύστημα. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιπαρατεθείτε σε ένα τέτοιο απαράδεκτο σύστημα. Ευχαριστώ και τελευταία στελικά ο κύριος Γιάρ. Uh, Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ερωτήσεις της συναδέλφου Μαγκίνε σε ό,τι αφορά τις ε, πληρωμές αυτές και πότε μπορούν να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις γιατί συνδέονται και με ένα κίνδυνο οι κυρώσεις να είναι πιο υψηλές από την ζημία. Θα γίνει λοιπόν διάλογος με τα κράτη-μέλη σε αυτή την πρώτη προγραμματική φάση γιατί Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις απάτης, δεν τις λαμβάνω υπόψη, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου γίνονται λάθη ε, χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόθεση. Μήπως θα συζητήσουμε λοιπόν τα μέλη. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις, ε, μισό λεπτό για την κάθε απάντηση. Έχετε 1,5 λεπτό, άντε το πολύ δύο, κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα, για να ε, ε, ελέγξουμε την ΕΦΑ, την, ε, το χώρο εστιασμένο στην οικολογία, αρκεί να έχουμε στο LPIS φωτογραφίες. Γι' αυτό προτείναμε και ένα τέτοιο στρώμα της ΕΦΑ. Τα κράτη-μέλη ζήτησαν αναβολή μέχρι το 2019. Ο κύριος Λαβίος, η ηγητή σας, συνέβαλε στο να μειώσουμε το χρόνο το 2018. Το 2018 τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να περιλάβουν στο ELPIS το επιπλέον στρώμα της ΕΦΑ. Αλλιώς, βέβαια, κάποιο κράτος που το επιθυμεί μπορεί να το ε, ε, επιβάλλει και νωρίτερα. Θα γίνει κυρίως με χάρτες ε, και θα υπάρξει για το ΕΦΑ 10% περισσότερη έλεγχη επιτόπου. Και το αργότερο μέχρι το 2018 θα χρησιμοποιείται το ELPIS ε, με πιο ευρύ και τεχνικά προηγμένο τρόπο. Κυρία Μόη, η ερώτηση σας ήταν πιο γενική και δεν είναι εύκολο να απαντήσω γιατί εμείς ε, εξετάζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και ειδικέ περιπτώσεις. Δεν μπορώ να σας δώσω μια γενική απάντηση. Από τη στιγμή που εντοπίζουμε ατασταλίες στις δαπάνες, είτε από το κράτος μέλος, είτε από το δικαιούχο, φυσικά αναλαμβάνουμε δράση. Κάνουμε τους ελέγχους Γνωρίζετε ότι και η ΟΛΑΦ επιλαμβάνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης και φυσικά αντλούμε και τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά συμπεράσματα. Στο παρελθόν είχαμε κάποιες δημοσιονομικές διορθώσεις στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο. Και άλλες χώρες, για να μην πω όλες οι χώρες μέλη, είχαν τέτοιες περιπτώσεις αδικαιολόγητων δαπανών ή παράνομων δαπανών στα πλαίσια της ΚΑΠ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι συγκεκριμένο κατά νου, μια ειδική περίπτωση, μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Η τρίτη ερώτηση υπευλήθη από τον κύριο Γιάρ. Θα ήθελα να διορθώσω την εντύπωση ότι η διαδικασία εκαθάρισης λογαριασμών είναι μια διαδικασία κυρώσεων όπου τα κράτη-μέλη πρέπει να επιστρέψουν περισσότερα από αυτά που αδικαιολόγητα δαπάνησαν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες ε, για να γίνει σωστός έλεγχος των λογαριασμών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δώσουν ε, ε, σαφή υπολογισμό. Και αξιολογούμε τον κίνδυνο με βάση ένα καταποκοπή ποσοστό, 2, 5 ή 10%. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως και από το δικαστήριο αυτός ο τρόπος υπολογισμού. Τώρα προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα δίνοντας συστηματικά τα κράτη-μέλη 20 δευτερόλεπτα μου έμειναν, δίνοντας συστηματικά στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να υπολογίσουν τον δημοσιονομικό κίνδυνο για το κονδύλιο σε ατομική βάση. Βέβαια, η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και κουραστική, αλλά είναι ο μόνος τρόπος που προβλέπεται πια από τον κανονισμό και είμαι πεπισμένος ότι χάρη στο νέο σύστημα θα σημειώσουμε και πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες, μισό, μισό λεπτό. Sorry, the second part of... Το δεύτερο τμήμα της ερώτησής μου δεν το απαντήσατε. Για τις κυρώσεις για το πρασινισμά. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε, δεν το ξέρω ότι είναι αργά. Ναι, λυπάμαι. Φυσικά το πρασίνισμα χωρίς τις κυρώσεις θα ήταν ένα εθελούσιο σύστημα. Χρειάζονται λοιπόν κυρώσει αν θέλουμε να είναι υποχρεωτικό το σύστημα του πρασινίσματο για τι πληρωμέ. Υπάρχει μια παραδοσιακή περίοδο όπου τα πράγματα είναι περίπλοκα και για του αγρότε και για τι κυβερνήσει. Γι' αυτό ο νομοθέτη αποφάσισε να μην επιβληθούν οποιασδήποτε κυρώσει τα πρώτα δύο χρόνια, μετά να περάσουμε σε κυρώσει 20% και να φτάσει αυτό τελικά σε ποσοστό 25% του ποσού πρασινίσματος. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης και στο τέλος του σεμιναρίου. Ε, δεν έχω κουράγιο να κάνω ανακεφαλαίωση γιατί είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Ο καθένας θα βγάλει μόνος τα συμπεράσματα. Πάντως εμείς έχουμε άμεση επαφή με τους αγρότες και ακούμε τους φόβους και τις ανησυχίες τους και ρόλος και καθήκον μας είναι να τους διαβιβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ληφθούν υπόψη. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερον, φοβάμαι ότι στην ακρόαση του προτινόμενου επιτρόπου ο άνθρωπος θα φοβηθεί και θα το βάλει στα πόδια, θα παραιτηθεί και δεν θα έχουμε ποιον να κάνουμε, ποιον να κάνουμε ακρόαση. Ελπίζω να μην είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα και πιστεύω ότι μετά την ακρόαση ο προτινόμενος επίτροπος θα δημιουργήσει μία να της κατάστασης. Πάντως οι περισσότερες ερωτήσεις έχουν χαρακτήρα περισυλλογής και όποιοι είναι χριστιανοί ξέρουν τι σημαίνει περισυλλογή. Έχουν ένα τέτοιο ευλαβικό χαρακτήρα περισυλλογής. Παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί μπορεί να ήμουν κάπως απότομος στα σχόλιά μου, κάπως όμως, αλλά... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήμασταν κοντά σχετικά στις ε, εκλογές και μερικοί θέλαν να πούνε μερικά σχόλια. Πάντως πιστεύω ότι παρά μερικές φορές κάποια σχόλια που ήταν κάπως σε, έντονο ύφο, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το σεμινάριο και κάναμε μια καλή προετοιμασία για τη μεταρρυθμίση αυτή, αλλά μερικές φορές θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Γιατί μερικές φορές επισημάνουμε κάποια πράγματα, αλλά ίσως δεν ήμασταν αρκετά αποφασιστικοί και θα πρέπει να επανέλθουμε σε ορισμένα από αυτά. Έχετε λάβει ε, τα συμπεράσματα των συντονιστών. Τις έχετε λάβει και γραπτός ε, τις αποφάσεις των συντονιστών ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 11.30 με 12.30 συνεδρίασαν σήμερα οι συντονιστές και αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις θα θεωρηθώ ότι εγκρίθηκαν οι αποφάσεις των συντονιστών. 6 και 7 Οκτωβρίου θα είναι η επόμενη συνεδρίαση των, των, της Επιτροπής μας για, το, για την 7η του μηνός δεν είναι σίγουρο, αλλά το 6 Οκτωβρίου σημειώστε το για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά τηρήσαμε τον χρόνο μας ή κάναμε κάποια υπέρβαση. Είχαμε μέχρι τις 6 ή μέχρι τις 6.30. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, λύεται η συνεδρίαση. Καλώς απόγευμα.